Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε με την απογευματινή μας συνεδρίαση. Το πρώτο μας θέμα είναι το σημείο 21 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, την κυρία Ρέιλι. Πρόκειται για την εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα εξαγωγικών πιστώσεων που τη χάνουν δημόσια στήριξης Έγιναν έρευνες για τις εξαγωγικές πιστώσεις των κρατών μελών και αυτό ήταν το πλαίσιο μετά από το οποίο βάλαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και πολύ χαίρομαι πραγματικά που είναι μαζί μας σήμερα η κυρία Ορέιλι και θα μας εξηγήσει, θα μας δώσει πληροφορίες και ενημέρωση για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα. και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτή η στήριξη εξαγωγικών πιστώσεων. Παρακαλώ κύριε Ρέιλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Λάγκε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως ξέρετε, η εντολή μου αφορά διοικητικά και όχι πολιτικά ζητήματα, οπότε η δουλειά μου δεν συμπίπτει με τι πολύ σημαντικέ αρμοδιότητε τη Επιτροπή σα. Όταν όμω αυτό συμβαίνει, συνήθω έχει να κάνει με το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συλλογή και ανάλυση συγκεκριμένων ε, ε, κατηγοριών πληροφοριών. Σήμερα θέλω να σα παρουσιάσω μια προσφυγή που έγινε στην υπηρεσία μου για το πώ διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αιτήσει ε, ε εκθέσει για τι φορεί εξαγωγικών πιστώσεων των 100 μελών. Είμαι στι τελευταίε φάσει τη σύνταξη τη έκθεση και σκοπεύω να κλείσω την υπόθεση σύντομα. Το Φεβρουάριο 2016 η ECAWATS, μια ένα διεθνή συνασπισμό ε, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών που παρακολουθεί του φορεί εκδοτικών πιστώσεων επέβαλε προσφυγή σε μένα. Οι φορεί αυτέ, όπως ξέρετε δίνουν οικονομική στήριξη σε εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε αγορές ε, λόγω χάρη σε αναπτυσσόμενε χώρε, που μπορούν να θεωρηθούν πολύ ρηψοκίνδυνε για τον κανονικό ιδιωτικό τομέα. Η προσφυγή ε, ε, ε γύρει ε, αμφιβολίε για τη συμφιλίωση τη οικονομική ανάπτυξη και τη ευημερία μαζί με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντο. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλουν αιτήσει εκθέσει για τα προγράμματα εξαγωγικών πιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Ευρωπαϊκού Νόμου. Βάσει αυτών των εθνικών εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει αιτήσει έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο που συμπεριλαμβάνει αποτίμηση των φορέων των εξαγωγικών πιστώσεων και το πώ συμμορφώνονται με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υποχρεώσει τη. Ο ενάγων αμφισβητούσε το κατά πόσον αυτές οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής είναι πλήρεις και ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος. Στη διεξαγωγή τη έρευνά μου γνώριζα τι ε, κρίσιμε παρατηρήσει τη Επιτροπή σα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα τον Ιούνιο του 2013, με εισηγητή τον κύριο Γιάννη Ξαντό. Αποφάσισα να διεξαγάγω την έρευνά μου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα με έρευνες από δύο ε, εθνικούς συναδέλφους μου, τον Ισπανό και Πολωνό ε, διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Δικτύου οι οποίοι έλεγξαν τι δικέ του εθνικέ κυβερνήσει και του φορεί του. Βάσει τη έρευνά μου, κατέληξα ότι η διαδικασία εκθέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιωθεί. Τα πορίσματα θεωρώ ότι συμπίπτουν με τι απόψει σα από την έκθεση του 2013. Στι 11 Μαου 2017, λοιπόν, ε, υπέβαλα τι εξή τρει προτάσει ε, προ ε, γνώση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητά με την ΕΕΔ και την Κοινωνία των Πολιτών και να εκδώσει μια αναθεωρημένη, ένα αναθεωρημένο κατάλογο δείγμα, τέμπλε για τα κάτι μέλη. Το νέο αυτό τέμπλε θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχέ από τι συνθήκε και τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με μια συγκεκριμένη φοβολογία για την καταγραφή μη οικονομικών θεμάτων. Δύο, βάσει των δεσμεύσεών τη ω προ το κάτι μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει κατευθυντήρε γραμμέ για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στο πώ ε, συμπληρώνουν τι εκθέσει του προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να βελτιώσει την διεξιδικότητα τη ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων. Τρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει μέτρα για να ενισχύσει την ανάλυση και αποτίμηση που ε, εφαρμόζει στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλει προ το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά πέριψε τι προτάσει μου, επιχειρηματολογώντα ότι αυτέ οι προτάσει ξεπερνούν το ε, ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εγώ διαφώνησα με αυτή την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στι 23 Μαου 2018 επανεξέδωσα την πρότασή μου ω ε, πλήρου ισχύω ε, συστάσει του διαμεσολαβητή. Τα συμπεράσματα μου βασίζονται σε τρει βασικέ παρατηρήσει. Πρώτον, ε, η διατύπωση του πρώτου παρατήματο του σχετικού κανονισμού 1233-2011 δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράγει επίση έκθεση για το Ευρωκοινοβούλιο βασιζόμενη στι πληροφορίε, περιλαμβάνοντα μια αποτίμηση που θα αφορά την συμμόρφωση με τι αρχέ των εξωτερικών εισαγωγικών πιστώσεων και του στόχου και υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εννοείται ότι συμπεριλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώ και στην προστασία του περιβάλλοντο. Δεύτερον, οι αρχέ τη ε, σωστή διαχείριση απαιτούν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προχωρούν σε αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να είναι ακριβή, αντικειμενική, ανεξάρτητη, διεξοδική και να βασίζεται στι κατάλληλε πληροφορίε. Εάν η νομοθεσία δεν προβλέπει ομοιόμορφα πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει περισσότερα από το ελάχιστο απαιτούμενο. Ε, χρειάζεται διεξοδική αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένου καταλόγου και σχετικέ ε, κατευθύνσει γραμμέ για τα κρατημέλη. Καταλαβαίνω ότι το Κοινοβούλιο στην έκθεση του 2013 ε, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση. Η ε, προσεκτική εξέταση των εκθέσεων της Επιτροπής από το 2011 έως 2004 δείχνει ήταν πάρα πολύ ε, κενές περιεχομένου και δεν βασίζονταν σε ανεξάρτητη και αντικειμενική ανάλυση και αποτίμηση. Για αυτού του λόγους κατέληξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαπράξει κακό διαχείριση Πρόσφατα έλαβα την τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ τι συστάσει μου. Η Επιτροπή υποστηρίζει, εμένει στην άποψή τη μάλλον, ότι ο κανονισμό δεν επιτρέπει να ε, πει προ τα κράτη-μέλη τι πληροφορίε θα πρέπει να τι παράσχουν. Όμω, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να αναλάβει μέτρα για να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολή εκθέσεων και να υλοποιήσει το περιεχόμενο των συστάσεών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα είπε ότι θα συζητήσει με το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον κατάλογο και το template και ε, την δυνατότητα να αλλάξει μεθοδολογία υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον, θα προτείνει ένα σχέδιο, αναθεωρημένο σχέδιο καταλόγου ε, σημείων προσυμπλήρωση, το σχετική ομάδα εργασία του Συμβουλίου και για τι εξαγωγικέ πιστώσει και την ΕΕΔ. Επιπλέον, θα διαβουλευτεί και με την κοινωνία των πολιτών. Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα ξαναδεί το θέμα αυτό στο μέλλον, εφόσον αναθεωρηθεί ο κανονισμό 1233-2011. Ενώ λοιπόν οι υποσχέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καλύπτουν όλε μου τι ανησυχίε, τουλάχιστον έχει γίνει ε, σημαντική πρόοδο. Ε, αναμένω την διαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και θα ξαναδώ τι εξελίξει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Μόλι χθε Έλαβα τα σχόλια των άγοντων ω προ την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ανάγων ε, έθεσε μια σειρά από σημεία. Ανησυχεί ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα συνεχίσει να αναλύει την συμμόρφωση χωρί να έχει τι απαραίτητε πληροφορίε για να ολοκληρώσει τέτοια είδου αξιολόγηση και επίση ότι τα κάτι μέλη θα πρέπει να γκρίνουν τον αναθεωρημένο κατάλογο ε, και το template προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δεν ανανεωθεί λοιπόν, ε, μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ο κανονισμό τη, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα θα αναλύσω τι τοποθετήσει και των δύο πλευρών και θα ολοκληρώσω την εξέταση τη υπόθεση του. σύντομα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Είμαστε διάθεσοι σα για ερωτήσει και απαντήσει. Τέλεια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ της διαμεσολαβήτριας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως ε, θα μπορούσε να μας εξηγήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εντοπίζονται τα προβλήματα. Δίτρου Σαμπάρτα από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις εξαγωγικές πιστώσεις που νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν την χάνει της ε, αναγκαίας προσοχής. Ναι, υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν αφορούσαν το περιεχόμενο της πολιτικής. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε πλήρως τη διαφάνεια στον τομέα της πολιτικής των εξαγωγικών πιστώσεων με ταυτόχρονο σεβασμό στις υποχρεώσεις και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που υπάρχει η διαφωνία είναι η ερμηνεία των ορίων που θεσπίζει ο κανονισμός όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διατύπωση του παραρτήματος 1 που παρέθεσε και η διαμεσολαβήτρια αναφέρθηκε στις τέσσερις μαγικές λέξεις «βάση των επαρκών πληροφοριών» και υπάρχει μια διάταξη στο παράρτημα 1 που ρητός ορίζει τι πρέπει να παρέχει το κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να παρέχει δεδομένα που σχετίζονται με, με περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, νέες δεσμεύσεις, κονδύλια και ε, όπου ε, υπάρχουν ε, ε συνδεόμενες ε, υποχρεώσεις. αυτό είναι το όριο, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τίθεται για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον κανονισμό. Επίσης, τα κράτη-μέλη καλούνται να περιγράφουν πώς λαμβάνονται υπόψη στις δράσεις τους τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτά. Στη βάση όλων αυτών των πληροφοριών, η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να διεξάγει την αξιολόγησή τη. Αλλά μα περιορίζει ο κανονισμό ω προ το πόσε πληροφορίε μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε νομική βάση στον κανονισμό για να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε. Εν τούτης, έχουμε λάβει πλήρως υπόψη μας κατά την ε, εκτέλεση των καθηκόντων μας, τις θέσεις του Κοινοβουλίου, το ψήφισμα, τι θέσει τη ε, κοινωνία των πολιτών, τι θέσει όπω αυτέ έχουν εκφραστεί από τα κράτη-μέλη. Όμω, μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαπιστώσει προθυμία να υπάρξει αναθεώρηση του καταλόγου ελέγχου. Όπω είπε και η Διαμεσολαβήτρια, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν τι εκθέσει του, κάποια συγκεκριμένη μορφή. Εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό checklist, αν θέλετε. Τα κράτη-μέλη και πάλι δεν θα ήταν υποχρεωμένα να τα ακολουθήσουν. καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος υποβολής εκθέσεων και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Γιατί μας ενδιαφέρει να γίνονται σεβαστοί οι στόχοι και οι υποχρεώσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής, επίσης, δεν έχουμε λάβει ποτέ καταγγελία παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου. Αλλά Εκτός εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει στο να καταρτήσουμε έναν αναθεωρημένο κατάλογο με, με έναν κατάλογο δεδομένων που θα υπερβαίνει τα όσα προβλέπει ο κανονισμός αυτή τη στιγμή, η, Κομισι... η Κομισιόν αυτή τη στιγμή έχει δεμένα τα χέρια της. Εμείς συμφωνούμε μαζί σας, συμφωνούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά μόνοι μας δυστυχώς δεν έχουμε την αρμοδιότητα να προχωρήσουμε σε όλα όσα μας ζητάτε. Άρα δεν είναι ένοχη η Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος. Η εισηγήτριά μας τι πιστεύει. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία διαμεσολαβήτρια ή διαμεσολαβητής, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι έχετε το καρτελάκι μπροστά σας που λέει διαμεσολαβητής, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Βγαίνουμε από μια διαπραγμάτευση η οποία κατέληξε θετικά για το θέμα των ξένων επενδύσεων και για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να φιλτράρονται οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται για την μεταφορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ ισχύουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε την υπόθεση αυτή, έχοντας υπόψη ότι οι διάφορες ε, εταιρείες αρμόδιες για τις εξαγωγικές ε, πιστώσεις πρέπει να περνούν από έλεγχο. Περνούν από την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία τους όμως πρέπει να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει αυτού λοιπόν ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις και στις διαπραγματεύσεις είναι σαφές ότι δεν είναι θέμα αρμοδιότητα συντονισμού των ε, εταιριών αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη αναθέτουμε ευθύνη και στις χώρες μέλη, αλλά βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επαληθεύουν, να ελέγχουν ότι αυτές οι υπηρεσίες οι εταιρείε ανταποκρίνονται και λειτουργούν βάσει των κανόνων που προβλέπονται. Είχαμε πέντε εκθέσεις και φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία κατέληγε κάθε φορά στο ίδιο συμπέρασμα. Και το υπογραμμίσατε κι εσείς. Δεν υπάρχει καταγγελία. Αυτό τι σημαίνει. Ότι τηρείται η συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως υπάρχει και το πνεύμα και το γράμμα του κανονισμού. Το πνεύμα των διαπραγματεύσεων ήταν ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει στις χώρες μέλη κατευθυντήριες γραμμές ώστε να τηρείται το δείγμα έκθεσης και βάσει αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει τις πληροφορίες και έτσι να μπορεί πιο εύκολα να ελέγξει ότι όντως γίνονται σεβαστές οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα κάθε φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του έχει εκφράσει την ε, δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και χαίρομαι που διάφορες οργανώσεις πήγαν στην με Διαμεσολαβήτρια και που κατέληξε σε τέτοια συμπεράσματα που έχει καταλήξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι δηλαδή δεν μας ικανοποιεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν δυσκολίες, έτσι. Οι διαπραγματεύσει ήταν σίγουρα δύσκολες, γιατί όταν ασχολείστε με την κοφάστε μέσα ή άλλους, προφανώς υπάρχει και θέμα εθνικής κυριαρχίας. Ναι, αλλά ακριβώ αυτό είναι που είναι δικιά σας ευθύνη. Είναι δικιά σας ευθύνη να φροντίσετε η Ευρωπαϊκή Εθνική Κυριαρχία να μην έρχεται σε αντίφαση με το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν μας λέτε ακόμα και σήμερα ότι περιμένετε από το Συμβούλιο να δείξει την καλή του θέληση ώστε ενδεχομένω να τροποποιηθεί ο κατάλογος κτλ. Συγγνώμη, εμείς δεν είναι αυτό που σας ζητάμε. Όπως λέει και η Ευρωπαίδια Μεσολαβήτρια, αυτό που σας ζητάμε είναι να δώσετε στο Συμβούλιο και τις κατευθυντήριες γραμμές και τον κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να γνωρίζουν για τις ε, υπηρεσίες τους που προχωρούν σε εξαγωγικές πιστώσεις. Χωρίς να τίθεται θέμα εθνικής κυριαρχίας. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και η Ευρωπαία Μεσολαβήτρια. Και ελπίζω, ελπίζω η Επιτροπή μας να αποφασίσει, να παρακολουθήσει τι θα γίνει στη συνέχεια. Επίσημα θα παρακολουθούμε την κατάσταση ώστε να υποχρέσουμε την Επιτροπή και μέσω της Επιτροπής της χώρες μέλη να τηρήσουν τον κανονισμό στον οποίο καταλήξαμε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να αντιδράσω κι εγώ, ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ σοβαρό και το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε εμπιστοσύνη ή όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ο κανονισμό, η οδηγία μάλλον 1233 του 11 που υποχρεώνει ετήσια να έχουμε στοιχεία για τους φορείς εξωτερικών πιστώσεων. Όμως, τελικά, δεν φαίνεται ότι ελέγχονται παρκώς οι φορείς αυτοί εξαγωγικών πιστώσεων. Η Ombudsman, η διαμεσολαβήτρια, ακριβώς καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία δεν δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως και πρόσφατα υπήρξαν πάλι επικρίσεις για τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη κατάσταση. Εμείς, και είναι ο ρόλος μας και το καθήκον μας, ο κοινοβουλευτικό έλεγχος. Συνεπώ, πρέπει να ελέγχουμε και ό,τι συμπεράσματα βγάλουμε να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Και όπως λέει και ο κύριο Ζαντό, πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά την υπόθεση συνέχεια. Πρόεδρος, μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μένα. θα συμβουλεύατε το Κοινοβούλιο να κάνει. Να ζητήσει τι, νέα αναθεώρηση της νομοθεσίας, τι, να στείλουμε επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο, να του πούμε ότι πρέπει κάτι να κάνει με τις χώρες μέλη. Τι θα μας συμβουλεύατε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί τώρα δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Και το είπατε και εσείς ίδια εξάλλου. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα σκεφτόμουν να, να πω εγώ στο Κοινοβούλιο πώς να συνεχίσει με την πολιτική του. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χώρες μέλη. Δεν έχουμε διαφωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πολιτική. Η διαφωνία είναι με το Συμβούλιο Δηλαδή εσείς θα υποβάλλετε αναθεώρηση της νομοθεσίας ώστε να έχουμε μια, κάτι, μια καλύτερη έκθεση. Η Επιτροπή πρέπει να δούμε η, κατά πόσο η αναθεώρηση μιας παραγράφου στο παράρτημα του κανονισμού είναι κάτι που θα ικανοποιούσε. Ξέρετε ότι μπορεί να υπάρξουν μεγαλύτερες αλλαγές που να χρειάζονται αναθεώρηση. Δεν αποκλείεται δηλαδή να γίνει αναθεώρηση του κανονισμού. Δεν το αποκλείουμε. Και τι λέει η διαμεσολαβήτρια από αυτού. Ναι, έχω διάφορα να πω. Ωραία, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσής μας για τα όρια του κανονισμού διαφωνούμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσετε. Μιλάτε για τη διατύπωση στο παράρτημα 1 ότι η Επιτροπή θα εκπονεί ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αξιολόγησης κτλ. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστείτε στο τα κριτήρια που θα λάβετε υπόψη σας για να εκπονήσετε την έκθεση αυτή. Βλέπετε, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η λογική. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ικανοποιητική αξιολόγηση. Αν εσείς λέτε ότι δεν έχετε αρκετές πληροφορίες για αυτήν και υπάρχουν κενά, εσείς λέτε ότι με τον κανονισμό μπορείτε να πιέσετε κάπως περισσότερο με κατευθυντήριες γραμμές και ένα αναθεωρημένο υπόδειγμα. Εντάξει. Πρόεδρος. Καλώς. Σίγουρα θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Είτε με ψήφισμα. Θα δούμε οι συντονιστές τι θα αποφασίσουν γι' αυτό. Πάντως η κατάσταση μετά από τρία χρόνια χωρίς ε, βελτίωση δεν είναι ικανοποιητική για μας πρέπει να τοποθετηθεί σαφώς στο Κοινοβούλιο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο έργο σας. So, next item is... Συνεχίζουμε. Επόμενο θέμα είναι ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας για τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που έχουμε για την εμπορική μας ατζέντα. Μετά το ατύχημα, πώς προχώρησαν ε, τα πράγματα με το σύμφωνο αυτό, τον Ιούλιο υπήρξε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στον Μπαγκλαντές και η Επίτροπος Μάλστρομ ήταν εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση για την τεχνική κατάσταση. Οπότε καλό είναι τώρα να συζητήσουμε για την κατάσταση. Πρέπει να συζητήσουμε τη συνέχεια, τους πάντων το μέλλον της συμφωνίας με μια συντονιστική ομάδα, να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε και μεγάλο κατάλογο αδυναμιών που παρατηρούνται όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Έχουμε και τον πρέσβη του Μπαγκλαντές μαζί μας για να το συζητήσουμε αυτό. Καλώς ήρθατε. Αρχίζουμε λοιπόν με τον πρέσβη. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση μετά στη Γενική Διεύθυνση Trade, Εμπορίου και μετά ε, στον εισηγητή μα. Παρακαλώ κύριε Πρέσβη για 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, για να συζητήσουμε για το πώς έχουν τα πράγματα και το πώς προχωρά το σύμφωνο βιωσιμότητας και το πώς ε, το βλέπουμε εμείς, πώς προχωρούν οι εργασίες ε, για την υλοποίησή του στο Μπαγκλαντές και κυρίως ως προς τη μεταφορά αρμοδιοτήτων βάσει του συμφώνου στις αρχές της χώρας. Η συμφωνία για τις κατασκευαστικές εταιρείες στο Μπαγκλαντές υπεγράφει το 2013 με ε, συμβολή ευρωπαϊκών εταιριών. Ήταν μια βασική συμφωνία μεταξύ μεγάλων εταιριών και λιανικών υποκαταστημάτων, υποκαταστημάτων τους μάλλον λιανικής, για να υπάρχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές θεωρεί ότι η βοήθεια που δόθηκε από διεθνείς εταίρους για να ενισχυθούν τα εργοστάσια που σκοπεύουν τις εξαγωγές ήταν πολύ σημαντική. Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι η συμφωνία είχε να κάνει με 1.500 με 1505 εργοστάσια ε, ε ένδυσης, πρέτα πορτέ, ε, και 900 εργοστάσια ε, για επεξεργασία. 91% είχε να κάνει με τις σχέσεις συνεργασίας, το 80% προέκυψε απευθείας από τη συμφωνία. Τα αργοστάσια ήταν περίπου αυτά που σας ανέφερα αριθμητικά και καλύφθηκαν ε, όσα ε, απέμεναν από την Εθνική Πρωτοβουλία. Για να υπάρχει ε, ε, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της, των εργασιών επισκευών και ε, αναδιαρρύθμισης ε, δημιουργήθηκε από το Μαγκλαντές η κυψέλη ε, σχετικής, της σχετικής δουλειάς, αυτό που ονομάζουμε εμείς DIFI, στη σχετική κρατική υπηρεσία. η κυψέλη αυτή συντονισμού, αυτό που ονομάζουμε εμείς RCC, τώρα ήδη λειτουργεί. ελέγχει και παρακολουθεί την πρόοδο του συγκεκριμένου προγράμματος της Εθνικής Πρωτοβουλίας και των εργοστασιών που αυτό καλύπτει και ασχολείται, έχει αναλάβει τις ευθύνες που προκύπτουν από τη Συμφωνία για να αξιολογήσει τα εργοστάσια και την πρόοδο που αυτά έχουν επιτελέσει στη μεταβατική τους περίοδο. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει αυξήσει το εργατικό δυναμικό και τα δημοσιονομικά κονδύλια τα τελευταία πέντε χρόνια για να ενισχύσει τις δυνατότητες της DIFE. Ε, ο προπολογισμό ε, του σχετικού τμήματος έχει πενταπλασιαστεί και σύνολο 679 θέσεων εργασίας έχουν δημιουργηθεί ε, οπότε η στελέχωση φτάνει τα χίλια άτομα. Επιπλέον, πέραν των ε, ήδη εργαζομένων μηχανικών που ασχολούνται με τις επισκευές, 60 ε, επιπλέον μηχανικοί ε, προσλήφθηκαν από την RCC για να διευκολύνουν αυτές τις εργασίες εξυγένσης αποκατάστασης. Επίση, άλλοι 57, ε, άλλοι μάλλον 7 μηχανικοί που έχουν να βοηθήσουν στην επιτάχυση των εργασιών, 6 θα ε, συμμετάσχουν και ακόμα περισσότεροι πολύ σύντομα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταβατικής Περίοδου το τελευταίο τρίμηνο του 2017 συνεργάστηκε με εκπροσώπους των κυβερνήσεων του εργατικού χώρου, των εργαζομένων και εργοστασιάρχες για να ε, μπορέσουν τα περισσότερα εργοστάσια να ακολουθήσουν τις επιταγές του RCC. Επίσης, οι εργοδότες, ο σύνδεσμος εργοδοτών του Μπαγκλαντές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα. Η προσφυγή ενός ε, ομίλου ε, που δικάστηκε από το το Δικαστήριο ε, τελικά απορρίφθηκε. ο Όμιλος θα πρέπει να φύγει από το Μογκλαντές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2018. Αυτή η μεταβατική λοιπόν συμφωνία θα λειτουργεί πολύ σύντομα βάσει του προγράμματος ε, παρακολούθησης της μετάβασης της κυβέρνησης και των συστάσεων εποπτείας της Επιτροπής για την παρακολούθηση της μετάβασης. Καταλαβαίνουμε ότι ακόρντε έχει προσφύγει και στο το Δικαστήριο του Μπαγκλαντές και υπάρχουν σχετικές συζητήσεις στη χώρα. Καταλαβαίνουμε, ελπίζουμε μάλλον ότι θα υπάρξει επιτυχής συμφωνία και μεταφορά των ορμοδοτητών προς την RCC. Ε, είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργοστασίων. Ε, στις αρχές της χρονιάς, τον Ιούνιο του 2018, το τέταρτο, η τέταρτη σύνοδος για το Σύμφωνο Βιωσιμότητας διοργανώθηκε εδώ στις Βρυξέλλες. Πήρε μέρος ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Υπουργός Εμπορίου του Μαγκλαντές. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μπαγκλαντές θα κοιτάξουν να βεβαιωθούν ότι υπάρχει υπευθυνότητα στη διαχείριση του όλου προγράμματος από τον κόσμο της βιομηχανίας και των εταιριών και ότι είναι ασφαλής η αλυσίδα παραγωγής. Όπως ε, συζητήθηκε στην τελευταία συνάντηση αναθεώρηση του Συμφώνου Βιωσιμότητα, ε, οι νόμοι εργατικοί του Μπαγκλαντές πρέπει να μεταρρυθμιστούν περαιτέρω ε, όπως προκύπτει από τα ανανεωμένα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Η Βουλή ε, του Μπαγκλαντές έχει περάσει ήδη τις σχετικές τροπολογίες στην νομοθεσία της και θα εκδοθεί σύντομα κυβερνητική απόφαση. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές συνεργάζεται στενά και με τον ILO, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, για να υπάρχει ένα πρόγραμμα βελτίωσης της απασχόλησης που θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Υπάρχει και διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρου για να βεβαιωθούμε ότι σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζεται το πρόγραμμα και για να δημιουργηθούν οι κρατικοί φορείς που απαιτούνται ώστε να υπάρξει σωστή υλοποίηση. Η κυβέρνηση του Μαγκλαντές συμφωνεί ότι αποζημίωση για τις ζημιές στον χώρο εργασίας ή τον θάνατο είναι θεμελιώδη δικαίωμα του κάθε Αλλά έχει τεράστιο κόστος όλο αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να υπάρξει ενίσχυση από όλους τους εμπλεκομένους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά στον βιομηχανικό μας κλάδο. Το Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης συνεργάζεται με, το, με τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις για να ε, μπορέσουν και οι δικοί τους ε, άνθρωποι να βοηθήσουν την όλη διαδικασία. Προβλέπουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα αποζημίωσης για εργασιακά ατυχήματα ή άλλα ε, για τον τομέα ένδυσης των Μπαγκλαντές. Θα βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζουμε τα διδάγματα της Συμφωνίας Αποζημιώσεων Ράνα Μπλάζα. Ε, και στο παρελθόν έχουμε πει ότι ο τομέα τη ένδυση και τα εργοστάσια ένδυση ε, παραγωγή ενδυμάτων στο Μπαγκλαντέ έχουν επιδοθεί σε ε, ε, εντατικέ εργασίε αποκατάσταση και εξηγήσει. Όμω, αν δούμε το τίμημα που έχει, έχουν καταβάλει για την παραγωγή του, τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Επίση, θέλουμε τη στήριξή σα για να παρουσιαστεί το Μπαγκλαντές ως πετυχημένο παράδειγμα στον παγκόσμιο χώρο του, της παραγωγής ενδυμάτων και για άλλες χώρες που παράγουν έτοιμα ενδύματα. Ιδίως στον τομέα της ασφάλειας του χώρου εργασίας. Το Μπαγκλαντές θα παραμείνει αφοσιωμένο στην επιδίωξη κοινών στόχων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις καλές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Σίλβριτς, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Καλησπέρα. Πρωτού σας δώσω κάποιες νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους ε, ευρωβουλευτές και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ για την υποστήριξή τους, τη συμμετοχή τους στην επικοδομητική σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με το σύμφωνο αυτό. Έχουμε την αίσθηση ότι συμφωνούμε στα περισσότερα και σημαντικότερα ζητήματα και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα υποστήριξης ε, για τους εταίρους μας στο Μπαγκλαντές. Όντως, όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, έγινε το τέταρτο, η τέταρτη συνάντηση υψηλού επίπεδου για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας, όπου είχαμε την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε σε υψηλό επίπεδο σημαντικά ζητήματα. Ε, όπως υπόθηκε ήταν ε, παρόντες ο Επίτροπος, ο Υπουργός Εργασίας. Η εικόνα που αποκομίσαμε είναι μεικτή. Στα θετικά το, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι το Μπαγκλαντές ε, καταβάλει συστηματικές και διαρκείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης ε, στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία, ε, τα εργασιακά δικαιώματα μέσω της σχετικής νομοθεσίας που θεσπίζεται. Θεσπίστηκε μια τριμερής διαδικασία διαβούλευσης, συλλογικών διαπραγματεύσεων, και μέσα προσφυγής για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις σοβαρές της ανησυχίες όσον αφορά την ανυπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί σε βασικά εργατικά δικαιώματα και ο Επίτροπος έχει ξεκαθαρίσει στην, ξεκαθάρισε στην ε, ε, συνάντηση ότι οι υποχρεώσεις του Μπαγκλαντές υπό τον ILO θα πρέπει να τηρηθούν συλλογικές διαπραγματεύσει, εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό και αξιοποιήσαμε την ευκαιρία της συνάντησης αυτής για να υπενθυμίσουμε στο Μπαγκλαντές τις ελλείψεις που υπάρχουν στην νομοθεσία της χώρας αλλά και την ελλειπή σε ορισμένε περιπτώσεις εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Χαιρόμαστε βεβαίως ότι τέθηκε σε ισχύ ε, ο νέος νόμος για τα εργασιακά Τον έχουμε λάβει, βεβαίως είναι στα ε, Πρέπει να περιμένουμε την μετάφραση για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του νόμου. Ε, πάντως, θετικό είναι το γεγονός ότι για να συσταθεί συνδικάτο σε ένα εργοστάσιο ε, απαιτείται πλέον μόλι το 20% των εργαζομένων. Πρόκειται για μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που προβλεπόταν με βάση τον παλαιότερο νόμο. Αυτό είναι θετικό και καλούμε το Μπαγκλαντές να κινηθεί ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση και να κατεβάσει το ποσοστό αυτό στο 10%. Επίσης, καλούμε το Μπαγκλαντές να καταργήσει όλες τις αντισυνδικαλιστικές προβλέψεις της νομοθεσίας, να επιτρέψει πλήρη ελευθερία ε, του συνδικαλισμού και να ε, ε, προτείνουμε επίσης το ε, Μπαγκλαντές να μειώσει τις περιπτώσεις απορρίψεων προσφυγών των συνδικάτων στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε όλες τις πρωτεβουλίες μας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουμε ενεργά σε όλες αυτές τις διαδικασίες και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δράσεις του Accord στο Μπαγκλαντές θα συνεχίσουν έως ότου η κυψέλη εξυγίανσης και εξορθολογισμού κριθεί ε, ικανή να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της χωρίς ε, εξωτερική βοήθεια. Πράγματι λοιπόν η Κομισιόν εξέφρασε τις, αν, τις ανησυχίες της σχετικά με, την το πρώιμο, τον πρώιμο τερματισμό των δράσεων του Accord. Επιμείναμε στο ότι το Accord πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Ελπίζουμε ότι έπειτα από την προσφυγή του Ακόρτ στο Ανώτατο Δικαστήριο το, η κυβέρνηση θα υποστηρίξει το Accord και θα συνεχίσει τις δραστηριότητες του στο Μπαγκλαντές. Σημειώσαμε και αυτό που είπε μόλις ο κύριος Πρέσβης, πώς οι διοικητικές ικανότητες της Κυψέλης ε, αυτής βελτιώθηκαν μεν, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει ε, να περιμένουμε και το, το αποτέλεσμα της απόφασης του εφετείου. Όλα αυτά που σας λέω τα έχουμε πει και σε άλλα φόρα. Το είπαμε και στην ομάδα 3 5 τον Οκτώβριο. Συμπεριλαμβάνονται και στην τελευταία έκθεση για την τεχνική κατάσταση που ε, δημοσιεύσαμε το Σεπτέμβριο του 2018. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τώρα. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για την πολιτική προσοχή που δίνει στο Μπαγκλαντές. Πρόσφατα μετά υπήρξε ψήφισμα ε, της 15ης Νοεμβρίου για αυτό το θέμα, αλλά συνεχίζετε να ενδιαφέρεστε, κάτι το οποίο μας βοηθά και εμάς πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέσεις από παλιά με τον Μπαγκλαντές και θέλω να υπογραμμίσω ότι η πολιτική μας δέσμευση έχει εντατικοποιηθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της προσφυγικής ε, κρίσης. Η κυρία Μογκερίνη συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Χασίνα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και με τον Πρωθυπουργό δύο φορές. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνει και η κυβέρνηση και ο κόσμος των Παγκλαντές για να υποδεχτεί τους Ροχίνγκα, τους πρόσφυγες, η πίεση είναι τεράστια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στο Μπαγκλαντές. Στόχος μας είναι βέβαια η επιστροφή των προσφύγων στις κατοικίε τους, αλλά αυτό πρέπει να γίνει βέβαια με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και εφόσον το θέλουν οι ίδιοι και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η κατάσταση βέβαια επίση στη Μιαμάρ πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή τους. Υπάρχουν πολιτικές δεσμεύσεις επίσης από το Πακιστάν για να εφαρμόσει τις ε, διαδικασίες που χρειάζονται για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι πρόσφυγες τα σπίτια τους. Όπως είπαμε βέβαια με αξιοπρέπεια. Εμείς περιμένουμε να συνεχίσει τη δέσμευσή του αυτή το Πακιστάν προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή όλες ε, οι σχετικές διατάξεις για να επιτευχθεί η επιστροφή των προσφύγων. Βλέπουμε θετικές εξελίξεις από πλευρά της κυβέρνησης πάντως και τη συμφωνεί με τον ΟΗΕ και γιατί ανταποκρίνεται στις δικές μας ανησυχίες. Υπάρχουν διπλωματικές διαβουλεύσεις που, ε, θα, που έγιναν μάλλον τον Ιούλιο στο Τακά και γενικά το Πακιστάν δείχνει ότι είναι διατεθμένο και έτοιμο να καλύψει τις αδυναμίες. Φυσικά η κατάσταση εξακολουθεί να μας ανησυχεί και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Πλησιάζουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει το διάλογο με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και το λέμε αυτό και στις διάφορες δηλώσεις μας. Η προετοιμασία τώρα των κοινοβουλευτικών εκλογών είναι κάτι που συζητάμε με τις αρχές της χώρας συχνά. Ε, περιμένουμε να, είναι, να γίνουν με διαφάνεια οι εκλογές αυτές, με τη συμμετοχή όλων, αναμερόληπτες, να υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε, προστασία του κόσμου κλπ. Η κυβέρνηση όντω θέλει την προστασία της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, κάποια μέτρα έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρέπει να εφαρμόσει πλήρως βέβαια τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας με ελευθερίες, συνδικαλιστικές και με το Μπαγκλαντές ακριβώς το συζητάμε αυτό το θέμα, το συζητάμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τακτικά στις διαβουλεύσεις μας. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Um, Mr. Carvin. Ευχαριστούμε, ο κύριος Κάρβιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μου είπατε πόσο χρόνο έχω. Οπότε, όπως θέλω. Σωστά. Καλά, εντάξει, ωραία, θα περιοριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ και εγώ τον πρέσβη και τα θεσμικά όργανα, τα ευρωπαϊκά, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Πρόεδρε, ειλικρινά, όσο μιλάω, τα σκέφτομαι αυτά που θέλω να πω, γιατί κοιτάξτε, ή πολύ εύκολα θα σας πω δύο λόγια και θα σας μεταφέρω ένα πολύ ισορροπημένο μήνυμα, το οποίο ε, θα βοηθήσει τον Μπαγκλαντές να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές και να το κάνουμε με πολύ διπλωματικό τρόπο. Η γλώσσα πάντως που χρησιμοποιείται από τους ευρωβουλευτές που με σταματούν στους διαδρόμους ε, μου εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπαγκλαντές. Αυτοί όμως η αντιμετώπιση είναι εντελώ διαφορετική από το ισορροπημένο μήνυμα που λάβαμε εδώ σήμερα. Φυσικά και καταλαβαίνω τη θέση την οποία βρίσκεται ο πρέσβης, καταλαβαίνω πολύ καλά επίσης την ε, θέση στην οποία βρίσκονται τα αδερφά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και γιατί σε αυτό εδώ το φόρουμ μεταφέρουν αυτά που μας μετέφεραν. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι οποίοι προσπαθούν να πετύχουν ισορροπία ανάμεσα στα όλο και πιο δύσκολα μηνύματα που μου φτάνουν από τους συναδέρφους και την εκτίμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα αδερφά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για παράδειγμα, σήμερα άκουσα την εξή φράση, ότι εξακολουθεί να είναι ανησυχητική κατάσταση και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Έτσι είπε η Ευρωπαϊκή Επίρρηση Εξωτερική Δράση. Πολλοί ευρωβουλευτέ ακριβώ αυτό λένε. Αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι ευρωβουλευτέ που έρχονται σε επαφή μαζί μου. Όπως και οι υπόλοιποι, και εγώ έχω πάρει αυτό το γραπτό για το τι θα πρέπει να πω σήμερα. Αλλά εγώ αντιστάθηκα δεν το είπα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο που πλέον θα πρέπει να είμαστε εντελώ ξεκάθαροι για το πού βρισκόμαστε. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προφανώς βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και απέναντι σε πολλά και διάφορα μέτωπα, όχι μόνο αυτό. Πάντως εγώ νομίζω ότι θα έχουμε πιο γρήγορα πρόοδο αν διατηρήσουμε τη γλώσσα της διπλωματίας. Και ειλικρινά το λέω. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αληθινή γλώσσα μέχρι να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει γρήγορα. Αλλιώς θα βλέπουμε κάποια κινητοποίηση εδώ στο σώμα που θα μπλοκάρει περισσότερο τα πράγματα και τις θετικές εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μπαγκλαντές. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ κρυφή γλώσσα, αλλά βλέπετε τι συμβαίνει στην περιοχή, στις γειτονικέ χώρες. Για καιρό λέγαμε και η Επιτροπή μας ότι πρέπει να υπάρχει περιθώριο για περισσότερο εμπόριο με το Μπαγκλαντές εξαιτία της κρίσης των Ροχίνγκα. Τώρα όμως οι συνάδελφοι τι λένε. Λένε καιρός είναι να αρχίσουμε να τοποθετούμαστε κανονικά πια. Αυτό μπορώ να πω. Φυσικά και θέλουμε να διασφαλίσουμε πρόσβαση σε όλα τα εμπορικά πακέτα, να προχωρήσουν και να μην πάμε πίσω. Αλλά για να γίνει αυτό πράγματι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις παρεμβάσεις που ακούσαμε. Άρα το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να δει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί τα λόγια από μόνα τους και κυρίως τα ωραία λόγια δεν φτάνουν πια. Ε, πρόεδρε, μου είπατε 5 λεπτά, 5 και 6 δευτερόλεπτα είναι. Τώρα σας απασχολεί ο συνάδελφο, αλλά τέλος πάντων δεν θα συνεχίσω περισσότερο, κάνοντας πώ δεν κατάλαβα ότι πέρασε η ώρα μου. Σας ευχαριστώ για αυτά τα πολύ ξεκάθαρα λόγια σας. Να δώσω το λόγο στην κυρία Λάμπερ, την επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσει με την Νότια Ασία. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι δεν είχα σκοπό να παρέμβω όμως θα πω ότι είναι εύλογες οι ανασυχίες που εκφράστηκαν. Τις έχουμε συζητήσει και εμείς με τον πρέσβη. Θέλω να τονίσω αυτό που υπόθηκε για την κρίση των Ροχίνγκα και το τι έχει γίνει ως προς την απορρόφηση, την υποδοχή ε, ικανοτήτων διοικητικού χαρακτήρα προκειμένου να ε, υπάρξει διαχείριση της κρίσης. Ξέρουμε ότι το Μπαγκλαντές έχει κατευθύνει πόρους προς την ε, διαχείριση της κρίσης αυτής και ξέρουμε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά την στήριξη που δόθηκε στον Μπαγκλαντές. Οπότε η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι είναι περίπλοκη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει κανείς να συνεκτιμήσει. Σχόλια για την εργατική νομοθεσία, για τις ζώνες εξαγωγών. Όλα αυτά που συζητούμε σήμερα είναι ζητήματα που μας απασχολούν εδώ και χρόνια. Τα έχουμε συζητήσει σε πολυάριθμες περιπτώσεις και με πολυάριθμες ευκαιρίες και σε επισκέψεις μας στη χώρα και βεβαίως πιστεύω και εγώ ότι η πρόοδος θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και ταχύτερη. Ε, και μας ανησυχεί επίσης η πρόοδος, ε, η κατάσταση γύρω από το Accord. Ξέρουμε επίσης ότι ένας σχετικά μικρός, αλλά παρόλα αυτά αριθμός ε, εργοστασίων ε, του Μπαγκλαντές το τελευταίο διάστημα έχει μειώσει τα περιβαλλοντικά του πρότυπα χωρίς να υπάρχει μείωση των τιμών ε, των προϊόντων. Γιατί πολύ συχνά ε, υπάρχει αυτή η συζήτηση του τι είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν. Εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία και μια ανισορροπία. Πρέπει και αυτή η διάσταση να ληφθεί υπόψη. Και βεβαίως, καθώς το Μπαγκλαντές ε, θα απομακρύνεται από, την, από το καθεστώς της ε, χαμηλής ανάπτυξης χώρας σε μεσαίας ανάπτυξης. Ε, αντιστοίχως βεβαίως ε, θα πρέπει και οι δικές μας προσδοκίες και απαιτήσει από το Μπαγκλαντές να αυξηθούν. Όλα αυτά θα έχουμε στην ευκαιρία και στην, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εμπορική συμφωνία με το Μπαγκλαντές να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θέλω να σας πω ότι οικονομικά τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ το Μπαγκλαντές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια τεχνική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα κείμενο το οποίο λέει πώς βρίσκεται το Πακιστάν σήμερα όσον αφορά την ε, σταθερότητα Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι για τα εργασιακά δικαιώματα. Το Μπαγκλαντές φαίνεται ότι συνεχίζει διευθυντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το εργασιακό δίκαιο. Και φαίνεται ότι θέλει να πετύχει και τις προδιαγραφές για το δικαίωμα του συνέρχεστε και συνδικαλίζεστε. Επίσης, δουλεύει και για τη βελτίωση των υποδομών, για τα κτίρια. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ακόρτ και επίσης να ξέρουμε πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα και στα δικαστήρια του Μπαγκλαντές. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που εξαρτώνται από το δικαστικό σύστημα και κινδυνεύουν να χάσουν πολλά παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το ότι οι αρχές του Μπαγκλαντές μπορούν να επιθεωρήσουν και να ελέγξουν όλη αυτή την κατάσταση, κατά πόσο δηλαδή όλα συνάδουν με το ακόρδι όχι. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ώστε το Μπαγκλαντές να τηρήσει όλα, όλες τις διατάξεις του ακόρδου. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Μπαγκλαντές πρέπει να πετύχουν συμφωνία με συνένεση ώστε οι αλλαγές να γίνουν με καλό τρόπο και να είναι βιώσιμες. Υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ακόμα, πολλά μένα γίνουν πράγματι και υπάρχουν και εκλογέ σύντομα. Κατά τη γνώμη μου, πολιτικά και στρατηγικά, Θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας χάρτης πορείας με συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό θα βοηθούσε την επόμενη κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ώστε να συμμορφωθεί προς ε, τα όσα προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Άγνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο κύριος Καρίμ, ούτε εγώ θέλω να κινδυνολογήσω, όμως ο χρόνος περνάει. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ε, ξεκινήσω έναν ε, συναγερμό, αλλά ο συναγερμός έχει ήδη αρχίσει να χτυπά από μόνος τους. Σε δέκα μέρες το ακόρι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα και παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος την προηγούμενη περίοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους της κλωστοϊφαντουργίας στο Μπαγκλαντές. Και με αφορμή την συζήτησή μας για την τεχνική κατάσταση, νομίζω ότι τα ευρήματα της έκθεσης αυτής είναι σαφέστατα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ε, ολοκληρωθεί το έργο του, του Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ε, έχει ε, συμφωνήσει να ολοκληρώσει το κορδ, το έργο του έως ότου η Κυψέλη ε, μπορέσει να αναλάβει εκείνη τα καθήκοντα αυτά, αυτό και είναι δεδομένο ότι οι κρατικές αρχές αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη τις ικανότητες και τις δυνατότητες να επιβάλλουν ε, τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στα εργαστάσια κλειστοφαντουργίας. Γι' αυτό και ε, καλέσαμε, η, κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μπαγκλαντές να δώσει μια μεταβατική περίοδο στο Ακόρντ και δυστυχώς πρέπει να πω ότι ο πρέσβης του Μπαγκλαντές δεν απάντησε σε αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο χρόνος περνάει. Γι' αυτό και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους ρωτώ πόσο σημαντική είναι για εσάς η λειτουργία του Ακόρντ για το Μπαγκλαντές και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας απέναντι στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί σε αυτή την συνάντηση υψηλού επίπεδου. Και φυσικά το ζήτημα δεν εξαντλείται μόνο στο θέμα του ακόρτ. Όμως το ερώτημά μου είναι, έχουμε 10 μέρες μπροστά μας. Τι θα κάνετε για να εμποδίσετε την εκδίωξη του ακόρτ από τη χώρα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό το σύμφωνο βιωσιμότητας έχει σαν στόχο να προστατεύει τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε δει τι γίνεται με την παγκοσμιοποίηση. Ε, όλο και μεγαλύτερη δύναμη έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι. Οι πολυεθνικές συγκεντρώνουν περισσότερη δύναμη, περισσότερα χρήματα. Και το αποκορύφωμα ήταν, για παράδειγμα, η φοβερή τραγωδία στο Ραζα Πλάζα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ξεφεύγουμε από τώρα και να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν δικαιώματα. Διαβάζουμε ότι η συμφωνία αυτή χρειάζεται άλλους έξι μήνες. Μα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσει αυτό το σύμφωνο βιωσιμότητας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Επίγει να απαιτήσουμε να προχωρήσει το σύμφωνο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν φτάνουν τα ευχολόγια. Ευχαριστώ. Θέλετε να αντιδράσετε, κύριε Πρέσβη. πολύ σύντομα σας παρακαλώ και αν γίνεται όχι διαβαστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε λίγο χρόνο για να απαντήσω σε ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ε, στην σημερινή συζήτηση. Όπως ε, δήλωσα και εισαγωγικά, και όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει η κυβέρνησή μου στο παρελθόν, θα πρέπει να έχουμε ένα πράγμα πολύ ξεκάθαρο. Το ακόρντ δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από τον Μπαγκλαντές. Υπήρξε μια συμφωνία για πέντε χρόνια με τον Μπαγκλαντές. Αυτή η περίοδος εκπνέει πλέον. Αυτό δεν έχει σχέση με καμία εκδίωξη. Και επιπλέον, ανέφερα ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του Ακόρντ, έχουν προσφύγει τα μέλη του Ακόρντ στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, η οποία και εξετάζεται και παράλληλα συνεχίζονται ανεπίσημες επαφές και συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Εμείς θέλουμε από τη διαδικασία αυτή να προκύψει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να είναι αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για τα άλλα ζητήματα που τέθηκαν. Για την πρόοδο την οποία σημείωσε ο κλάδος και τον Μπαγκλαντές. Ξέρετε ότι ο κλάδος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μου. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε γρήγορες λύσεις. Φυσικά θα πρέπει να είναι όσο πιο πρακτικές γίνεται οι, λύσεις που επιδιώκουμε. Αλλά δεν μπορούν να δοθούν γρήγορες βιαστικές λύσεις σε έναν τόσο κρίσιμη σημασίας κλάδο για τον Μπαγκλαντές όπως είναι η κλωστοϊφαντουργία. Πριν από 40 χρόνια εξαρτιόμασταν ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό από την βοήθεια που μας παρήχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν λέω ότι όλη αυτή η βοήθεια έχει πλέον υποκατασταθεί από το εμπόριο, όμως βρίσκεται σε μια διαδικασία, αν θέλετε, υποκατάστασης, σταδιακής αντικατάστασης της βοήθειας με εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό έχει αποτελέσει και πρότυπο για άλλες χώρες παραγωγής έτοιμου ενδύματος, με τις οποίες βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία και με τις οποίες έχουμε φιλικότατες σχέσεις. Τα λέω αυτά ως προς τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Κομισιόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν επίσης έχει ξεκαθαρίσει στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει συγκεκριμένα και μακρόπνοα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ιδίω τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων προκειμένου να μπορούμε να αιτιολογήσουμε την συνέχιση των, των, της συνεργασίας μας μέσω του πρωτοσμησιακού καθεστώτος που παρέχουμε στα προϊόντα του Μπαγκλαντές. Το λέω αυτό για να γνωρίζουν όλοι ότι υπό αυτήν την ενισχυμένη εμπλοκή, συμμετοχή, διοργανώσαμε και μια αποστολή, επίσκεψη το Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της οποίας βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της ανάλυσης τους. Θα καταλήξουμε όμως σε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση και η έκθεση που θα συντάξουμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα συμπεριληφθεί και θα ληφθεί υπόψη στα επόμενα βήματα που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Αλλά και εμείς συμμετέχουμε εδώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παροτρύνουμε τον Μπαγκλαντές να σημειώσει απτή πρόοδο. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Στηρίζουμε και την ΑΚΟΡΤ για όσα έχει προσφέρει στον Μπαγκλαντές και στην βιομηχανία ένδυσης εκεί και συνεχίζουμε τις σχετικές συζητήσεις μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων. Ωραία. Ολοκληρώνουμε και με αυτό το σημείο θα θυμόμαστε την πολύ σαφή τοποθέτηση του εισηγητή μας. Είναι ζήτημα που επήγει. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ωραία. Περνάμε στο 23. Τριμερείς διάλογοι. Δεν έχουμε πολλά να πούμε, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ένας τριμερείς διάλογος. Ο λόγος των υπεύθυνων της επιτυχίας, τον κύριο Προύστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια καλή είδηση να σας ανακοινώσω. Πριν από μία ώρα μόλις, οδηγηθήκαμε σε θετικό αποτέλεσμα σε τριμερή διάλογο, στον τριμερή διάλογο για το μηχανισμό των ξένων επενδύσεων, τον, τη μέθοδο ε, διήθησης, φιλτραρίσματος Ξέρετε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο σωστού φιλτραρίσματο των ξένων επενδύσεων, που δεν έχει σκοπό να τι περιορίσει, αλλά να είμαστε πιο ε, ξεκάθαροι ω προ τι περίεργε επενδύσει. Αυτέ που δεν ανταποκρίνονται σε, σε οικονομικέ σκοπιμότητε, αλλά πολιτικέ. Εδώ και 1,5 χρόνο υπήρχε μια έκθεση πρωτοβουλία που ήταν. Ε, ε, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, επειδή μια σειρά από κράτη, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, αποφάσισαν να επιληφθούν, ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεση, κάτι που δέχτηκε ο κ. Γιονκέρ πολύ γρήγορα. Και μετά εργαστήκαμε συστηματικά και μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο τον Νοέμβριο. Ήταν πολύ σημαντικό να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα τώρα και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μπέρντ Λάγκε, τον πρόεδρο, ο οποίος με βοήθησε ιδιαίτερα στι διαπραγματεύσει. Διαπραγματεύσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Ήταν ε, σημαντικό να πάμε γρήγορα, διότι σήμερα ο κόσμος της οικονομίας προχωρά πολύ γρήγορα και περιμέναμε την έκθεση αυτή για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εργαστήκαμε λοιπόν με πολύ γοργό ρυθμό αλλά και με πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν ε, κοιτάξαμε να βιαστούμε και να έχουμε χειρότερο περιεχόμενο. Ίσα ίσα θελήσαμε να ενισχύσουμε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής συμπεριλαμβάνοντας ένα τρίτο σενάριο, το χειρότερο δυνατό σενάριο, όταν ένα κάτω μέλο δίνει μια αρνητική τοποθέτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, αποφανθεί. Δεν ήταν κάτι που ήταν σαφές πώς θα επιληθεί. Επίσης για τα πεδία αρμοδιοτήτων πετύχαμε να τα διακρίνουμε σωστά, έχοντας ένα σύνολο τομέων που καλύπτονται, ε, που αφορούν ε, από τη δημόσια ασφάλεια και τάξη μέχρι ένα σωρό άλλα θέματα και διατηρήσαμε τον στόχο του πραγματισμού και της αποτελεσματικότητας. Δεν ε, δημιουργήσαμε νομίζω ένα περιττό νομοθέτημα, αλλά κάτι που θα χρησιμεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Και πιστέψτε με, ήταν ε, πραγματικό κατόρθωμα όλο αυτό, γιατί πριν από ένα χρόνο πολύ λίγα κρατημέλη επιθυμούσαν αυτή την ε, μέθοδο δίθησης, φιλτραρίσματος. Και όπως έλεγε και ο συνονόματός μου, ο Μαρσέλ Προύστ, ήμασταν στην αναζήτηση του χρόνου που έχει χαθεί ε, με την ε, προσπάθεια αυτή. Ήταν απαραίτητο το εργαλείο ε, φιλτραρίσματο των ξένων επενδύσεων, γιατί το έχουν όλοι οι υπόλοιποι διεθνεί παράγοντε εκτό από εμά, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη λοιπόν είναι μια αγορά ελεγχόμενη, υπό Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Αφού αρνηθήκαμε την, ε, ε, το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, μετά την απόρριψη του TTIP, επιτέλους δείξαμε ότι πάψαμε να είμαστε αφελείς ως Ευρωπαίοι με αυτό το τρίτο βήμα. Πολύ καλή δουλειά αυτή που κάναμε. Προωθήσαμε τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Congratulations. I think Ευχαριστώ συγχαρητήρια. Το Κοινοβούλιο νομίζω πέτυχε ένα καλό αποτέλεσμα και μάλιστα εντάχει. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος τρομερής διάλογος. Κανονισμός των ε, εγγύησεων. Όπως θα ξέρετε, κάθε εμπορική συμφωνία συνοδεύεται από κανονισμό εγγύησεων. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν οριζόντιο τέτοιο κανονισμό για όλε τι εμπορικέ συμφωνίε. Όπω έγινε με την Νότια Κορέα, την Κολομβία, το Περού και το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό. θα ισχύει για, για την επόμενη γενιά συμφωνιών μας με την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Τριμερής διάλογος λοιπόν έχει ξεκινήσει επί Αυστριακή Προεδρία χθε μόλι. Οι διαπραγματεύσεις χωρίστηκαν σε τρία σύνολα και τρεις υποομάδες ώστε να μπορούν να συζητηθούν πολλά διαφορετικά σημεία εν παραλίλω. Ο εξυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποτιμησή της, τεχνικές τροπολογίες για την επικαιροποίηση του TDI, και κάποια άλλα ήταν σημεία στα οποία επετεύχθη πρόοδος και πότε οι περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου έγιναν αποδεκτές από τα άλλα θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και κάποια σχέδια κειμένου για τις συμβαστικές. Απογοητευτικό για το Κοινοβούλιο ήταν ότι για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα σχετικά σημεία δεν υποβλήθηκε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι μάλλον ακατανόητο, διότι στον κανονισμό μας σε όλους τους κανονισμούς εγγύσεων, έχουμε κάποια αποκτή παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το εμπόριο με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό στις συμφωνίες με την Κολομβία, το Περού, την, ε, το Εκουαδόρ, γενικώ στην Νοτιοαμερική ας πούμε. Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Αυστρική Προεδρία δεν δέχτηκαν τι τροπολογίε μα, δεν έγινε καμία συμβαστική πρόταση λοιπόν. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει χθε την όλη συζήτηση για τον οριζόντιο κανονισμό. Τώρα θα ξαναβρεθούμε στις 28 Νοεμβρίου και ίσως να πετύχουμε κάποια πρόοδο. Ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 24. As you... Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε αντιπροσωπεία μας στη Χιλή, όπου να είναι. Τελευταία πριν τα Χριστούγεννα αποστολή μας εκεί για να δούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της εμπορικής μας συμφωνίας με την Χιλή. Θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα, θα προετοιμάσουμε κάπως δηλαδή τις συζητήσεις που θα κάνουμε στα τέλη Δεκεμβρίου στη Χιλή. Γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ματίας Γιόγκερσον ο οποίος είναι υπεύθυνο και του δίνω το λόγο ευθύ αμέσω από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, δηλαδή για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι κάπως ως καιρός τώρα που δεν σας έχουμε μιλήσει για τη χιλή. Θα ήθελα να μπορώ να σας παρουσιάσω περισσότερη πρόοδο από ό,τι έχει πραγματικά επιτευχθεί μέχρι σήμερα αλλά σας ενημερώνω, σας προειδοποιώ ότι πρόκειται για διαπραγματεύσεις πολύ σημαντικές, αλλά που δεν έχουν προχωρήσει όσο γρήγορα ή όσο πολύ θα θέλαμε. Ποιο είναι το πλαίσιο. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις το Νοέμβριο πέρυσι. Ξεκίνησε τότε η διαδικασία διαπραγματευσεις τον νοεμβριο περυσι ξεκινησε τοτε η διαδικασια δηλαδη με έναν πρώτο γύρο και τον Ιανουάριο είχαμε άλλον έναν πολύ ουσιώδη και άλλον έναν ουσιώδη γύρο ε, συνομιλιών είχαμε το Μάιο. Επετέχθη πρόοδος, μπορέσαμε μάλιστα και να θέσουμε όλες τις αρχικές προτάσεις μας ε, στο τραπέζι, είχαμε και τις προτάσεις της Χιλής, ακούσαμε και τις δικές τους δηλαδή, οπότε βλέπετε ότι σε αυτούς τους ε, γύρους προχωρήσαμε ικανοποιητικά. Όμως, είναι σαφές ότι υπάρχουν ε, τομείς, κάποιοι λίγοι, όπου είναι πιο δύσκολο να προχωρήσουμε ε, με την χιλή σε σχέση με αυτό που προσδοκούσαμε. Ακριβώς γιατί αναλύουμε με λεπτομέρειες ε, τα ζητήματα. Για κάποια από αυτά δεν θέλησε η χιλή να προχωρήσει όπως είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις, όπως είναι οι επενδύσεις, η διαιτησία δηλαδή για τους επενδυτές, η προστασία των επενδύσεων, το IPR, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως επίσης και οι πρώτες ύλες. Από τον Ιούνιο που μας πέρασε, προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε και για αυτά τα ζητήματα. Είμαστε σε επαφή με τη Χιλή για να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είχαμε κάποιες συναντήσεις, επαφές πιο σωστά, η Επίτροπος με τον ε, ομόλογο που άλλαξε στο μεταξύ στη Χιλή. Και έγινε και μία συνάντηση με τον πρόεδρο Γιούγκερ και τον πρόεδρο Πινιέρα τον Οκτώβριο. Προς το παρόν θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο να προχωρήσουμε και κυρίως για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Αλλά επίσης και για την πρόσβαση στις αγορές. Εμείς θέλουμε να τα συζητήσουμε αυτά. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε έναν επόμενο γύρο που προβλέπεται για τον Ιανουάριο. Βέβαια πρέπει να το επιβεβαιώσει η Χιλή. Στη Χιλή θα γίνει αυτός ο γύρος συνομιλιών. Οπότε εξαρτώμαστε από την προθυμία και από την πρόσκληση βέβαια των χιλιανών. Συνολικά πάντως εμείς θέλουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές γιατί έτσι εξυγχρονίζεται η συμφωνία αυτή έχει ξεπεραστεί αρκετά, δεν υπάρχει ρήτρα βιωσιμότητα μέσα. Θέλουμε να ξεχρονίσουμε λοιπόν και αυτή τη συμφωνία με τη Χιλή. Και διμερός είναι πολύ σημαντική συμφωνία και θα ήταν καλό να στείλουμε ένα μήνυμα με τη Χιλή ότι είμαστε υπέρ του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες. Αυτές είναι οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Τέλεια. Πάνω στην ώρα ήρθε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτικής Δράσης. Γνωρίζετε ότι υπάρχει και συμφωνία σύνδεσης η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο, δεν συζητούμε δηλαδή μόνο για τον εξυγχρονισμό της εμπορικής συμφωνίας. Για τρία λεπτά θα μας μιλήσει ο κύριος Καστενουίτα για την Συμφωνία Σύνδεσης. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που μόλις κατέφθασα. Μιλάμε για τη χιλή, φαντάζομαι. Ε? Ναι. Διαπραγματευόμαστε εδώ και ακριβώς ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε στις 16 Νοεμβρίου του 2017. Έχουμε κάνει αρκετά σημαντική ικανοποιητική πρόοδο στα πολιτικά θέματα οι χιλιανοί εταίροι μας έχουν επιδείξει και επικοδομητική στάση και ευελιξία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά αποζητήματα. Τη μη διάδοση, τη μετανάστευση, την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και έχουμε ήδη ολοκληρώσει συζήτηση για 38 άρθρα τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στην εντολή μας και νομίζω ότι απομένουν μόλις 11 άρθρα. Κάτι που δείχνει ότι έχουμε ολοκληρώσει ήδη το 75% του κειμένου που είχαμε ε, να συζητήσουμε με τους ε, ε, χιλιανούς. Από αυτή την άποψη είμαστε ικανοποιημένοι. Τα εναπομείνατα ζητήματα, κάποια από αυτά βεβαίως είναι δύσκολα, φορολογία, μη διάδοση, θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση που θα εξασφαλίζει τα ενωσιακά συμφέροντα, όμως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Χιλή είναι πρόθυμη στο να προχωρήσει τον εξοχρονισμό της συμφωνίας και να ανοίξει νέους τομείς συνεργασία και πολιτικού διαλόγου. Είναι πλέον μια χώρα μέσου εισοδήματο και από αυτή την άποψη είμαστε εταίροι σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ε, αντιμετωπίζουμε και τις ίδιες προκλήσεις απέναντι ε, σε τρίτες χώρες. Δεν έχουμε συζητήσει ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα της συμφωνίας μας, γιατί αυτό συνδέεται με τα όσα συζητούμε στο κεφάλαιο για το εμπόριο, καθώς και κάποια άλλα οικονομικής φύσεως ζητήματα. είναι ζητήματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί η συζήτηση στην εμπορική συμφωνία για να δούμε πώ θα τα διαμορφώσουμε σε αυτή τη συμφωνία που σα περιγράφω εγώ. Δεν προβλέπεται να γίνει κάποιο επίσημος γύρος αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση, γιατί περιμένουμε να δούμε ποιε θα είναι οι εξελίξει στι συζητήσει για την εμπορική συμφωνία. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζονται κανονικά οι τεχνικέ ανταλλαγέ απόψεων. Κάνουμε και βίντεο διασκέψει που επίση μα επιτρέπουν να σημειώνουμε πρόοδο επί του κειμένου που μα υπέβαλαν τα κράτη-μέλη προκειμένου να συζητήσουμε με την ε, Χιλή. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί, ταυτόχρονα όμω διατηρούμε και τον ρεαλισμό μα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφωνίε στο, το, στον τομέα του εμπορίου και εκεί θα πρέπει να επιδείξουμε υπομονή έω ότου καταλήξουμε στι τελικέ φάσει τη διαπραγματεύση. Θα χρειαστούμε το μεγαλύτερο μέρο του 2019 για να συνεχίσουμε τι συζητήσει, όμως σε, συνεδρίαση που είχα σήμερα το πρωί με τα κράτη-μέλη εκφράστηκε η πεποίθηση και η ελπίδα ότι το έργο αυτό θα στεφθεί εντός του 2009 με, 10, ε, με επιτυχία. Πρόεδρος, ναι, το 2019 φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εμπορικές συμφωνίες. Λοιπόν, η συγκίτριά μας είναι... Η Ήμα Πινιέρο. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ τους εκπροσώπους της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θέλω να καλωσορίσω και τον πρέσβη τη Χιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συνεργάτες του που τον συνοδεύουν. Πρώτα απ' όλα, θέλω να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει ο εξυγχρονισμός αυτής της συμφωνίας. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι. Συμφωνία που, όπως είπε και ο κύριος Γιόγκερσεν, είναι από τις αρχές του αιώνα που πρέπει να εξυγχρονιστεί. Θέλουμε να δώσουμε διαφορετική, διαφορετικό βάρος σε αυτές τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή ήταν εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονταν και από τις δύο πλευρές και φαίνεται ότι χάνουμε πολλές ευκαιρίες στις εμπορικές μας σχέσεις. Γι' αυτό και οι συμφωνίες αυτές είναι ξεπερασμένες και θέλουν εξυγχρονισμό. Όμως εμένα με απασχολεί πολύ το πανόραμα που έχουμε μπροστά μα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ελπίζαμε ότι σε αυτήν την ε, θητεία με αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Μπορεί να λέγαμε, εντάξει θα ήταν ίσως δύσκολο, αλλά θα ήταν εφικτό. Τώρα όμως έχουμε απογοητευτεί. πάντα στις διαπραγματεύσεις προκύπτουν κάποιες δυσκολίες τεχνικής φύσεως στο περιεχόμενο. Μένα όμως με ανησυχεί πολύ γιατί έχουμε τέτοια καθυστέρηση, για ποιο λόγο υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τις τεχνικής φύσεως δυσκολίες. Όταν υπάρχουν ε, δυσκολίες για μια συγκεκριμένη πτυχή μπορούμε να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες πτυχές. Εδώ όμως από πλευρά της Επιτροπής έχουν δημοσιευθεί 18 κείμενα προτάσεων η, Κύλη, η Χίλη συγγνώμη, έχει δημοσιεύσει 8 περιμένουμε στα τέλη Ιανουαρίου κανονικά την σχετική έκθεση. Φαίνεται ότι υπήρξε ένας πρώτος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών τον Μάιο που μας πέρασε για να συζητηθεί ο ξυγχρονισμός της συμφωνίας και έγινε και διάλογος και τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο ώστε να ετοιμαστεί με την κοινωνία των πολιτών ε, η πρώτη εκδοχή του Συμφώνου Βιωσιμότητας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία και εμείς πάντα λέγαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο. Οπότε η διαπραγματευτική ομάδα συνεχίζει ίδια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής εκτός από τον επικεφαλής Οπότε έχει συμφωνηθεί η προοπτική, το πλαίσιο εφαρμογής. Οπότε θα ήθελα να καταλάβω περισσότερο και περισσότερο σε βάθος ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε στις διάφορες πτυχές της συμφωνίας. Έπειτα πιστεύω και υποστηρίζω ότι δεν θα πρέπει να πέσει καθόλου η φιλοδοξία μας για τη συμφωνία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πρόσβαση στις αγορές, τις γεωγραφικές ενδείξεις, το σύστημα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι ζητήματα σημαντικά, όπως και η προστασία των επενδύσεων. Όταν είχα την ευκαιρία να πάω στη Χιλή, και είχαμε και την επίσκεψη των βουλευτών της Γερουσίας και του Κογκρέσου που συνόδευαν τον πρόεδρο Πινέρα στις Βρυξέλλες, συναντηθήκαμε και δεν γνωρίζουμε καλά το μοντέλο, το σύστημα δηλαδή διαιτησίας για τις επενδύσεις. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το γνωρίζουμε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Οπότε μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτού του είδους την ε, διαπαιδαγώγηση, δηλαδή να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Το σύστημα του ISDS ε, λειτουργήσε καλά καταρχήν. Σήμερα υπάρχουν 17 συμφωνίες επενδύσεων με τις χώρες μέλη που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αλλά είναι θέμα γνώσης και να συνειδητοποιήσουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να στηρίξει επίλυση ε, διαιτησία που να επαφίεται σε ιδιωτικούς φορείς. Γι' αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χιλή επίσης. Γιατί δεν θα έπρεπε αυτό το στοιχείο να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε. Και ολοκληρώνουμε μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα των ποσοστώσεων των προτιμησιακών Είμαστε στο 95-96% τα τελευταία χρόνια με τη Χιλή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι 75%. Δεν μπορεί να αυξηθεί αυτό το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα καλέσω τον ε, Προεδρευτή της Χιλής να σχολιάσει για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο ταξίδι σας στη Χιλή. Να είναι καρποφόρα η διαμονή σας εκεί και να ευχαριστηθείτε την ε, χώρα μας και να καταλάβετε και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την ανάπτυξή μας. Επιβεβαιώνω τη βούλησή μας και τη δέσμευσή μας υπέρ των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα. Πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάτι σημαντικό να φτάσουμε σε αναβάθμιση της ε, σημερινής συμφωνίας. Είναι μια δέσμευση την οποία επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Χιλής που ήταν εδώ τον Οκτώβριο και μίλησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ. Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου και είμαι αισιόδοξο και για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους διαφωνούμε. Αλλά Υπάρχει μια μεθοδολογία. Σε αυτήν πρέπει να συμφωνήσουμε για να προχωρήσουμε. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Όχι μόνο στο πολιτικό σκέλος και τις συνεργασίες, αλλά και στο εμπορικό σκέλος. Έχουμε σημαντικά αποτελέσματα ήδη. Και ελπίζω σύντομα να προχωρήσουμε περισσότερο και στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, όπου δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε καταλάβει πολύ καλά. Γνωρίζουμε τι είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις και βασιζόμαστε σε αυτές για τα αλκοολούχα ποτά, τον ίνο. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς αυτήν την έννοια θα τη συμπεριλάβουμε στην εμπορική συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Εμείς δεν είμαστε κατά των γεωγραφικών ενδείξεων. Καθ' άλλο. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία διευρύνεται με το trademark. Συνεχίζω πάντως να παρακολουθώ ε, τη συζήτηση. Θα υπάρξει ένας νέος ο γύρος και εμείς είμαστε ανοιχτοί για τον γύρο αυτό. Όπου ελπίζουμε να έχουμε την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών. Ένα χρόνο έχουν συμπληρώσει οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι πολύ. Άλλες φορές είναι δύο χρόνια παραπάνω. Ωραία, καλά θα ήταν να ήταν πιο σύντομα τα αποτελέσματα. Αλλά τι να κάνουμε, κάθε διαπραγμάτευση έχει τη δικιά της δυναμική. Ελπίζω στην επόμενη χρονιά να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό επιθυμούμε, αυτό θέλουμε. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες μας. Ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ματίας, ε, πολύ θετικά ακούγονται τα πράγματα από όσα μας είπε μόλις ο πρέσβης. Τα δικά σχόλια ποια είναι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο πρέσβης. Υπάρχει μεγάλη προσήλωση και από τις δύο πλευρές και αυτό επικυρώθηκε και στη συνάντηση Πινιέρα Γιούγκερ τον Οκτώβριο. Θέλω όμως ε, να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Πινιέρου. Ότι δεν πρέπει να μειώσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου. Διότι πρώτον έχουμε εξαιρετικές εμπορικές σχέσεις με τη Χιλή και έχουμε μια ολοκληρωμένη ήδη συμφωνία. Η όποια αναβάθμιση λοιπόν θα πρέπει να υπερβαίνει τα σημερινά όρια, να αποτελεί πραγματική αναβάθμιση και να μας δώσει ε, έμπνευση για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να ε, μπορούμε να εξηγήσουμε την όποια απόφαση πάρουμε και στους εσωτερικούς ε, εμπλεκόμενους μας, ε, τα κράτη-μέλη στη δική μας περίπτωση. Αυτή η διαδικασία βεβαίως είναι χρονοβόρα, αλλά είναι αναγκαία για να υπάρχει υποστήριξη όλων των πλευρών. Υπάρχουν λοιπόν οι δυνατότητε για να επιτύχουμε ένα καλό επιτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, ευαισθησίε των ε, δύο πλευρών. Κατανοώ πλήρω αυτά που είπε ο πρέσβης. Ε, θα συζητηθεί και μια ανταλλαγή ως προς την πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά με τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με την Χιλή είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Τέλεια, λέει ο Πρόεδρος. E η Ευρωπαϊκή ε, ε, Υπηρεσία Εξωτικής Δράσης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ακόμη και αν η δική μας ε, δουλειά είναι λίγο διαφορετική, πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας. Ε, το έχουμε συζητήσει πολλάκις και με ε, τους ευρωβουλευτές. Έχουμε ήδη επιτυχεί αρκετά, ακριβώς γιατί υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τη Χιλή, μια συμφωνία ε, γύρω από μια σειρά αποζητήματα, αλλά παρόλα όσα συνέβησαν και τις αλλαγές που θα υπάρξουν εδώ στο Κοινοβούλιο, είμαστε ε, γεμάτη ελπίδα ότι του χρόνου θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις δύο διαδικασίες για τη Συμφωνία Σύνδεση και την Εμπορική Συμφωνία. Ο κύριος Σταρμπάτη. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μπροστά μου ένα κείμενο. Και θα διαβάσω την παρέμβασή μου. Είναι σαφές ότι η διαδικασία εξυγχρονισμού σκοπό έχει να αξιοποιήσει το δυναμικό στις διμερείς ε, συναλλαγές και ανταλλαγές αγαθών που είχε ευθύνουσα τάση το 2017 και 2018. Πρέπει να είμαστε φιλοδοξότεροι και να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία στον εμπορικό πυλώνα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ενέργεια, συγκεκριμένου τομεί ε, για τις μικρομεσαίες και τις μικροεπιχειρήσεις, τις δημόσιες προμήθειε. Επίσης, ένα ενιαίο σύνολο για τις επενδύσεις, για να αντικαταστήσουμε τις συνθήκες δημερών επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μάλλον αρκετών κρατών μελών και της Χιλής και να επιδιώξουμε το νέο μοντέλο για την επιθυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αλλάζει ε, το σύστημα επίλυσης διαφορών ISDS με ένα σύστημα που βασίζεται στο κρατικό δικαστικό. Τις αναφέρουμε τις προτάσεις αυτές στην έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας του Ιουλίου 2017. Οι συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους τρεις διαγματευτικούς γύρους πώς τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είναι δύσκολο και πού θα σκοντάψει όλη η διαδικασία. Ποιο είναι το γεωπολιτικό πλαίσιο η Χιλή δεσμεύεται για την απελευθέρωση του εμπορίου ανέκαθεν. Έχει ε, 22 εμπορικέ συμφωνίε με πολλέ χώρε που καλύπτουν την Κίνα, την Ινδία, τον Νότιο Κορέα, το Μεξικό, τη Μερκοσούρ και το καθεξή. Είναι η πρώτη Αμερικανική χώρα που πήρε μέρο στον ε, ΠΟΕ. Έχει οικονομική ανάπτυξη το 2018 με 0,8% και έχει υπογράψει συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία με σκοπό να ε, τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2018 πώς εντάσσονται οι δικές μας διαπραγματεύσεις σε αυτή την ευρύτερη εικόνα και πώς θα προοδεύσουμε στις σχετικές συνομιλίες. Εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στη Χιλή, ζητήματα που εδώ και καιρό δεν έχουν επιληθεί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάπως. Συνάδελφοι μου ανέφεραν συγκεκριμένα κεφάλαιο όπως την ισότητα των φύλων ή τα μέτρα για τη μη συμμόρφωση. Έχουν συζητηθεί κάποια αυτά προκαταρτικά με του εταίρου μα και ποιε είναι οι ποτέ του αντιδράσει. Ήταν η παρέμβαση τη κυρία Μακλάρη. Εντάξει, τα καταγράφουμε. Θα τα ρωτήσουμε και στην επίσκεψή μα στο τέλο Δεκεμβρίου. Είμα. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θέλουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Αλλά συγχρόνως πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεμπλοκάρουμε τα θέματα αυτά τα οποία δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, ο κύριος Γιόγκερσεν μπορεί να μου απαντήσει για τα προτιμησιακά ποσοστά, τα επίπεδα δηλαδή προτιμήσεων. Και ο πρέσβης μπορεί να μας πει εμείς που θα πάμε στη Χιλή ε, τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη βοήθεια για τις διαπραγματεύσεις αυτές, ώστε να προχωρήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Τέλος, ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μακλάρκιν, που τις παρατηρήσεις της θα τις λάβουμε υπόψη. Πρόεδρος, έχει να σε βουλέψει τίποτα ο πρέσβης? Πρόεδρε, το μόνο που θα μπορούσε που θα μπορούσα να τολμήσω να προτείνω στην Εμακουλάδα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Χιλή. Δεν τολμάω να κάνω προτάσεις γιατί γνωρίζει τη χώρα πάρα πολύ καλά. Έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σε πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το εξή. Η Ευρώπη αποτελεί σημείο αναφορά για τη Χιλή. Ένα σημείο αναφορά όχι μόνο γιατί είναι ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο, αλλά επειδή είμαστε πολύ κοντά σε θέματα αξιών και αρχών, που είναι κοινέ μεταξύ μα. Δεν είναι ρητορική αυτό, είναι κάτι ουσιαστικό στην σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη Χιλή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να το επαναλάβουμε και στη Χιλή, όχι μόνο εδώ. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είσαστε μια προστιθέμενη αξία, ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Χιλής. Μπορεί να μην είναι ο πρώτος, έχουμε άλλους δύο που είναι πιο σημαντικοί, αλλά εσείς είσαστε μια πρόσθετη αξία για μας. Γιατί έχετε μια ολοκλήρωση, εκπροσωπείτε διάφορες αξίες και αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κράτος δικαίου και στις πρακτικές σας και τις πολιτικές σας τις εμπορικές. Είσαστε λοιπόν προστιθέμενη αξία και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο και εμείς δουλεύουμε για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας Σύνθεσης, τόσο τον πολιτικό πυλώνα όσο και τον εμπορικό και τα δύο σκέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πεπισμένοι ότι όλα αυτά θα συζητηθούν ενδελεχώς κατά την επίσκεψή μας που θα πιούμε πολύ καλό κρασί από τη Χιλή. Άλλα σχόλια, ναι, μια πολύ σύντομη απάντηση στην κυρία Ροντρίγκη Πινιέρο για τον βαθμό απορρόφησης. Ε, είναι αλήθεια για την Χιλή και για τις ευρωπαϊκές εταιρείε δεν είναι κάτι που είναι συνηθιστό, είναι κάτι που το βλέπουμε σε αρκετέ συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους μας όπου οι δεσμολογικές προτιμήσεις που έχουμε προσφέρει με τις συμφωνίες μας κινητοποιούν τις εταιρείε μας. Είναι δύσκολο να πούμε ότι υπάρχει ένας και μόνο λόγος γι' αυτό, αλλά πιστεύω είναι ότι μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν αρκετά για το θέμα. Το εξετάζουμε λοιπόν αυτό ως κατάσταση, όχι μόνο ως προς τη χειλή, αλλά και άλλες συμφωνίες. Περισσότερη δουλειά μπορεί να γίνει για την προσφορά περισσότερων πληροφοριών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίω είναι και ρόλο των κρατών μελών να κάνουν κάτι γι' αυτό. ώστε οι εταιρείε να αξιοποιούν τις δυνατότητες που ε, μπορούμε να πετύχουμε εμείς με τις εμπορικές μας συμφωνίες. Δική του αρμοδιότητα είναι η πραγωγή των ε, εξαγωγών τους με τους σχετικούς φορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε το σημείο 24. Ευχαριστούμε τον πρεσβευτή τη Χιλής που ήρθε από την πρεσβεία του και περνάμε στο 25. Αυτό το σήμερα το απόγευμα έχουμε όλη τη Λατινική Αμερική. Περνάμε στο Μεξικό. Και θα μιλήσουμε για την εμπορική συμφωνία και τη σύναψή τη μετά την επίσκεψη συγκέντρωση στοιχείων που έγινε τον Ιούνιο στο Μεξικό. Νέα ναύτα προβλέπεται. Ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις μας με, τη, με το Μεξικό. Κύριε Γιόγκερσεν, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είπατε τόσα πολλά με μία φράση. Ανακεφαλαιώνοντας. Μεξικό. Για να μην μακρηγορήσω. Ξεκινήσαμε το 2016. Πετύχαμε πρόοδο, ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε εντατικέ διαπραγματεύσει, ολοκληρώθηκαν φέτο, τον Απρίλιο του 2018 και το αποτέλεσμα ήταν φιλόδοξο και διεξοδικό. Πολύ καλή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Επιτρόπου Εμπορίου, της Επιτροπής δηλαδή, και της κυβέρνησης του Μεξικού. Με τη συμμετοχή του κ. Γουαχάρδο, του Υπουργού Οικονομικών. Οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν σωστά και τι πρέπει να κάνουμε για να δημοσιευτεί το κείμενο είναι αυτό που μένει. Όπως ξέρετε έχουμε δημοσιεύσει και άλλα κείμενα στο παρελθόν. Από τις διακοπές του καλοκαιριού εργαζόμαστε εντατικά σε συνδυασμό με το Μεξικό για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την τελευταία εκδοχή του κειμένου και του σχετικού πληροφοριακού υλικού και ε, κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος. Τις επόμενες ημέρες ελπίζουμε ότι θα δημοσιεύσουμε τα κείμενα που δεν έχουν δημοσιευτεί για τους κανόνες προέλευσης, για τα προ... προϊόντα, για τις ε, διευκόλυνσεις ε, τις εμπορικές, για τα πνευματικά δικαιώματα, για τη διοικητική συνεργασία, για τα αυτοκίνητα, το κεφάλαιο για τα εμπόρια και αγαθά, τα σχετικά πρωτόκολλα και παραρτήματα και επίσης πρέπει να δημοσιεύσουμε και τα προγράμματα πρόσβασης για την αγορά για τα ε, γεωργικά και τις ζωοτροφές και τις σχετικές υπηρεσίες. Όλα αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα. Και όλα αυτά για σκοπούς διαφάνειας σε συνεργασία με το Μεξικό. Τα δημοσιεύουμε εν παραλίλω, ταυτόχρονα. Τα ίδια κείμενα. Επόμενα βήματα. Νομική με επιμέλεια των κειμένων και από τις δύο πλευρές, διότι αυτό που θέλουμε είναι όσο δυνατόν συντομότερα να ολοκληρώσουμε με τις επίσημες εργασίες και να υποβάλουμε τις προτάσεις για να υπογραφούν. Το μόνο που μένει να γίνει επί της ουσίας είναι να συμπληρωθεί το παράρτημα για τις δημόσιες προμήθειες σε υπομοσπονδιακό επίπεδο το Μεξικό δημοσιεύτηκε να το κάνει αυτός μέρος της πολιτικής συμφωνίας. Και αυτό θα είναι μέρος της τελικής συμφωνίας που προτείνουμε και σε εσά για να την εγκρίνετε. Ελπίζουμε στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς να έχουμε ολοκληρώσει. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση του Μεξικού και τις εκπροσώπους της ε, στενά και θα συνεχίσουμε αφού αναλάβει και η νέα κυβέρνηση του Μεξικού την 1η Δεκεμβρίου. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν θα παρακολύσει την ταχεία διεξαγωγή των διπλωματεύσεων. Ε, bring ε, forward as rapidly as possible the, ε, the former proposals for signature. Όσο το δυνατόν συντομότερα θα σας επιβάλλουμε επίσημες προτάσεις προς υπογραφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συζητήσαμε και τη Συμφωνία σύνδεση. Καλό λοιπόν την ΕΙΕΔ, τον κύριο Φερνάντο Πόντς αυτή τη στιγμή να μα πει τι γίνεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο, διότι ο Ματίας τα είπε όλα. Σας έκανε μια πολύ καλή επισκόπηση του πώ έχουν τα πράγματα. Η συμφωνία καλύπτει και πολιτικέ εξέλιξει και τη σχετική συνεργασία και εμπορικά. Είναι συμφωνία σφαιρική, εξυγχρονισμένη με έναν από του στρατηγικού μα εταίρου. οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα εξυγχρονιστεί και επικαιροποιηθεί ε, προ όφελο και των δύο πλευρών. Επί τη αρχής ξέρετε ότι συμφωνήσαμε και για τα πολιτικά και εμπορικά από το τέλος του 2017 Ακολούθησε συμφωνία για τα πολιτικά αρχέ τη αρχέ τη φθηνή χρονιά και από τι δύο πλευρέ, Μεξικού και Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται προσπάθειε να οδηγηθούμε γρήγορα σε αίσιο πέρα. Μόλι ολοκληρωθεί το κείμενο, κάτι που θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να κλείσουν και οι διοικητικέ διαδικασίε, θα γίνει και η νομική επιμέλεια, κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει. Από το τέλος των δημοκρατήσεων κιόλα θα γίνουν οι μεταφράσεις, οι οποίες θα χρειαστούν λίγο χρόνο, αλλά μετά τη μετάφραση η συμφωνία θα αποσταλεί αμέσω στο Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο αποφασή του Συμβουλίου Προσέγγιση, και μετά το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συμφωνή γνώμη του, συγγνώμη, ε, αφού μελετήσει τη συμφωνία. Εάν δοθεί και σύμφωνη γνώμη, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία από αυτή την πλευρά τουλάχιστον. Μετά και η διαδικασία κύρωση βεβαίω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τα κάτι μέλη. Δημοσίευση και ούτω καθεξής. Συγχαίρουμε τους εαυτούς μας. Καμαρώνουμε. Και συγχαίρουμε και τους Μεξικανούς συνεργάτες μας τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Λίγες είναι διατάξει που παραμένουν ακόμη προ συζήτηση. Θα πάψω. Αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Η φράση κλειδί σήμερα από την Κομισιόν και την ΕΕΔ είναι το «Είμαστε πολύ κοντά». Τη χρησιμοποιήσατε πολλέ φορέ σήμερα στι συζητήσει που είχαμε. Είμαστε πολύ κοντά. Ήρμα, εσύ πόσο κοντά είσαι. Bueno, yo también lo llevo hace tiempo, pero también... Και εγώ το λέω εδώ και καιρό. Η πρόβλεψη ήταν ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα είχαν τελειώσει όλες οι τεχνικές πτυχές. Τώρα και πάλι με τη μετάφραση, την αναθεώρηση των κειμένων κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περισσότερο χρόνο. Θυμάμαι ότι στην Επιτροπή μας πάντα εγκρίναμε μια τροπολογία ώστε η Γενική Διεύθυνση Trade να μπορεί να έχει στη διάθεσή της το προσωπικό ε, και γενικά ότι πόρους χρειάζεται για να ανταποκρίνεται στις προθεσμίες, αλλά δεν κερδίζουμε ποτέ στην Ολομέλεια. Τώρα για τη συμφωνία με το Μεξικό. Εγώ είμαι υπέρ τη δουλειά που έχει γίνει, που αποτελεί ένα καλό παράδειγμα πώς μπορούμε γρήγορα και ικανοποιητικά να εργαζόμαστε. Γιατί ανάμεσα στη συμφωνία που υπήρχε και αυτή στην οποία καταλήγουμε, υπάρχει ένα γιγάντιο βήμα και όσον αφορά το περιεχόμενο, το βάθος, αλλά έχουν συμπεριληφθεί και νέες καινοτόμε πτυχές που έχουμε για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κεφάλαιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα συγκεκριμένο ε, σημείο επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι πολύ βασικό σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Έπειτα έχει διευρυνθεί η πρόσβαση στην ε, αγορά. 340 γεωγραφικές ενδείξεις έχουν εγκριθεί. Οπότε έχει υπάρξει αλλαγή στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων, αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Πάντως και το Μεξικό έκανε τεράστια προσπάθεια. Η αηφόρος ανάπτυξη τώρα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι επίσης κάτι καινούριο που παλιά δεν είχε καμία συμφωνία. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο κεφάλαιο που μιλάει για την τήρηση των στόχων για το 2030, για την βιωσιμότητα, το περιβάλλον, την κοινωνική διάσταση και τα εργασιακά. Θέλω να συγχαρώ το Μεξικό που ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση 98. Ήταν μία από τις 8 που ήταν σε κρεμότητα. Οπότε πιστεύω ότι έχει κάνει εκπληκτική δουλειά το Μεξικό. Το μόνο που με θλίβει είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο για τη διάσταση του φύλου. Και έχω να κάνω μια πρόταση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Μεξικό έχουν υπογράψει στον Buenos Aires την δήλωση για τη διάσταση του φύλου. Είναι τόσο δύσκολο να ενσωματωθεί σε μια συμφωνία σύνδεσης. Μα δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε το 50% του κόσμου απ' έξω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για τη διαφάνεια. Σήμερα μπορείς να δεις τις προτάσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους, τα διάφορα δελτία με τις πληροφορίες. Δεν ισχύει όμως το ίδιο ε, με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αποτελείται μια συμφωνία από τρεις πυλώνες και το Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών μόνο στον εμπορικό πυλώνα έχει πρόσβαση δεν ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά την συνεργασία και το πολιτικό σκέλος. Οπότε μπράβο στο Μεξικό για την διαφάνεια με την οποία δούλεψε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ισχυώδεις μας δυστυχώς ε, είναι στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΒ αυτή τη στιγμή και μιλούν σήμερα για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό και μου ζήτησε να σας μεταφέρω δύο πτυχές της ε, συμφωνίας ε, που σχετίζονται και με αυτά που μόλις είπε η Μακουλάδα. Πιστεύει λοιπόν ότι οι ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή είναι ανυπαρκή ανεπαρκές, ανεπαρκής και εμείς διαφωνούμε και με, την, με το ενδεχόμενο να ενταχθεί ένα ICS στη συμφωνία. Πρόκειται για το σύστημα ε, διαμισολεύησης, για τις επενδύσεις που δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές να πλήττουν ε, τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ, γιατί θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με την ΑΚΤΑΚ, το Μεξικό είναι από τις πιο, πιο ε, διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο. Έχει μάλιστα αναγκαστεί από διεθνή δικαστήρια να καταβάλει τεράστια ποσά, 246 εκατομμύρια, σε επενδυτές. Αυτά δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο για το Μεξικό, αλλά και για άλλες περιοχές του κόσμου. Το Μεξικό, λοιπόν, ε, αντιμετωπίζει πλέον ε, τον κίνδυνο να ε, δεχθεί μηνύσει από ευρωπαίου επενδυτέ, αλλά και αντίστροφα. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως η Ισπανία μπορεί να δεχθούν τέτοιες μηνύσει από επενδυτές και να κληθούν να καταβάλουν τεράστια ποσά. Ε, αναφέρομαι και στον ε, Μεγιστάνα Κάρολ Στριμ, ο οποίος επιδίδεται ε, επιμακρών και συστηματικά σε τέτοιου είδου διαδικασίες. Δεύτερον Πιστεύουμε ότι η συμφωνία δεν είναι επαρκής όσον αφορά την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τήρησή τους από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένε υποχρεώσεις δεσμευτικού χαρακτήρα, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανισορροπία των συνεργασιών προκειμένου να προστατευτούν τα κέρδη. Σταματώ εδώ. Θα μπορούσα να σας δώσω και περισσότερα παραδείγματα που έχει συλλέξει η Λόλα. Αλλά έχω και εγώ ένα τρίτο ερώτημα. Ο κανονισμός για το ελάχιστο εισόδημα και η νέα συμφωνία είπα Καναδά και Μεξικό θα μπορούσε να οδηγήσει την αυτοκινητοβιομηχανία στο Μεξικό να μπει σε μια φθήνουσα πορεία, γιατί δεν είναι ανταγωνιστική έναντι των ε, αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Τι σημαίνει αυτό για μας. Δεν θα πρέπει και εμείς να εισάγουμε ένα θέμα που σχετίζεται έναν κανόνα για, την, ε, για το ελάχιστο εισόδημα των εργαζομένων. Κάτι τέτοιο θα ήταν συμμετρικό από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβανομένου υπόψη του τι έχει συμφωνηθεί από το Μεξικό με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Ευχαριστώ πολύ. Η, Κομισιόν. Για την ερώτηση της κυρίας Ροντρίγκε, αν υπήρξαν αλλαγές στα όσα έχουν συμφωνηθεί τον Απρίλιο, στις γεωγραφικές ενδείξεις για παράδειγμα. Όχι, δεν έχουν υπάρξει αλλαγές. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συμφωνία, μια πολύ φιλόδοξη συμφωνία και τόσο το Μεξικό όσο και εμείς είμαστε πολύ διεξοδικοί και θέλουμε να σημειώσουμε την ταχύτερη δυνατή πρόοδο. εξετάσαμε μια σειρά από θέματα, αλλά η διαδικασία αυτή πλέον έχει ολοκληρωθεί. Θα δημοσιευθούν τα σχετικά στοιχεία, θα τα δείτε κι εσείς τις επόμενες μέρες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω λοιπόν. Υπήρξε πολιτική συμφωνία και θα δημοσιευθούν όλα τα στοιχεία στα οποία ε, έχουμε καταλήξει το συντομότερο δυνατό και προσβλέπουμε πλέον στην ε, συνεργασία μας με την κυβέρνηση της χώρας για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Δεύτερον, για τα σχόλια του κυρίου Σόλτς. Έχετε τις απόψεις σας για το ICS. Εμείς διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε το πώς το σύστημα ε, δικαστηρίων για τις επενδύσεις θεωρούμε ότι είναι καλύτερο από ε, Πολλέ ε, επενδυτικέ συμφωνίε τι οποίε έχουν συνάψει τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει διεξοδικά και επιμακρών με το Κοινοβούλιο. Άλλωστε, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συμφωνία με τον Καναδά. Εμεί έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα διαιτησία που προτείνουμε. Είναι πιο διαφανές, περιλαμβάνει περισσότερα εχέγγυα και εξασφαλίσεις, περιορίζει τις δυνατότητες κατάχρησης ε, των νομικών μέσων. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε κίνδυνο οι εταιρείε να προσφεύγουν καταχρηστικά και διαρκώς εναντίον κρατών. Για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι ένα θέμα που σας απασχολεί και εσάς και εμάς. Είναι ένα θέμα που σίγουρα αφορά το Μεξικό, τη μεξικανική κοινωνία, τη μεξικανική κυβέρνηση γίνονται προσπάθειε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς από πλευράς εμπορική συμφωνίας είναι να ε, δώσουμε στους εαυτούς μας, εαυτούς μας περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να βοηθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση της εξελίξη στο Μεξικό και θα δείτε ότι αυτά που έχουμε συμπεριλάβει που δεν υπάρχουν ε, στην ισχύουσα συμφωνία, δηλαδή το κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, νομίζω ότι πλέον η νέα συμφωνία μας δίνει καλύτερα εργαλεία από αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα στα χέρια μας, αλλά είναι και γενικό το ερώτημα αυτό που καλύτερα θα ήταν να απαντήσει η ΑΕΔ. Για τον ελάχιστο μισθό δεν έχουμε ελάχιστο μισθό ούτε καν εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να πάμε Δηλαδή και να καθορίσουμε κάτι τέτοιο σε εμπορική συμφωνία με άλλη χώρα νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετικά τολμηρή κίνηση την οποία εμείς επιλέξαμε να μην κάνουμε. Πρόεδρος, και για την συμφωνία Ευρωπαϊκής, ε, είπα Μεξικού Καναδά, UMSCA, όταν εγκρίθηκε η USMCA, ε, εμείς βεβαίως είχαμε κάποιες ανησυχίες για το ότι θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και αντίκτυπο στην ε, συμφωνία που εμείς είχαμε συνάψει με το Μεξικό. Η ανάλυση μας όμως είναι ότι εν τέλει δεν αλλάζει με τίποτα και σε τίποτα τα όσα έχουν συμφωνηθεί με το Μεξικό αυτό άλλωστε ήταν και η προσδοκία μας από το Μεξικό που θεωρούμε ότι είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και προς τα εκεί ε, έτειναν άλλωστε και οι εγγύησει που λαμβάναμε από την κυβέρνηση του Μεξικού Για τις γεωγραφικές ενδείξεις για παράδειγμα, στον, ένα τομέα στον οποίο έχουμε επιτύχει πολλά, εκεί τα πράγματα είναι πλήρω εξασφαλισμένα ω προ το τι έχουμε κάνει εμεί και τι έχουμε συμφωνήσει εμεί με το Μεξικό. Βεβαίω υπάρχουν ε, μεγάλε διαφορέ όσον αφορά του τους, ε, ε κανόνε για την ε, προέλευση ανάμεσα στη δική μας συμφωνία με το Μεξικό και την συμφωνία του Μεξικό με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα καταλήξει να, ε, σε εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πίσω πόρτας. Αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να επηρεάσει, να επηρεάσει αρνητικά πιθανές ε, επενδύσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο Μεξικό. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ζυγίσει και να το σταθμίσει το Μεξικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πόνς, διαφάνεια λοιπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Ματίας και να υπογραμμίσω ότι η νέα συμφωνία πράγματι περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο πολλές. Έχει βεβαίως ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βασίζεται στις τελευταίες εξελίξεις αλλά ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να εντάξουμε και ουσιώδεις διατάξεις όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιγράφουμε με ποιον τρόπο ακριβώς οι δύο πλευρές θα συνεργάζονται για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στο Μεξικό όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί αυτό είναι το πνεύμα που διαπνέει τη συμφωνία. Πρόκειται για αμοιβέ δεσμεύσει. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει όσον αφορά τη διακήρυξη του Buenos Aires για τις προτάσεις που ακούστηκαν εδώ στην αίθουσα, ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε πολύ προηγμένο στάδιο της διαδικασίας πλέον. Είμαστε, σχεδόν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Ε, εναπομένουν πολύ λίγες διατάξει που βρίσκονται υπό συζήτηση πλέον. Αυτό όμω που μπορώ να σα πω είναι ότι αυτά που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμή συνιστούν ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα μα δώσει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μα συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του φύλου που και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν εν τέλει από την πολιτική βούληση να αξιοποιηθούν αυτέ οι διατάξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παρόλα αυτά οι διατάξει υπάρχουν, έχουν κατοχυρηθεί ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά, γιατί όπως είπατε και εσείς δεν υπήρχε εντολή. Έχουμε όμως πλέον τα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά, αν θέλετε. Το μόνο που θα απαιτηθεί βεβαίως θα είναι η πολιτική βούληση και αυτό μένει να αποδειχθεί αν θα υπάρξει. Θέλω επίση να συγχαρώ την συγγήτρια για το εξαιρετικό της έργο. Πράγματι, η πρακτική δημοσίευσης των ε, κειμένων διαφέρει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όσον αφορά αυτό που κάνει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τα κείμενα τα οποία είναι, για τα οποία είναι υπεύθυνη η υπηρεσία εξωτερική δράση. Αυτό είναι ένα γεγονό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Μεξικό. Είναι μια γενικευμένη πρακτική με την οποία μπορεί κανείς να συμφωνεί περισσότερο ή λιγότερο, αλλά πάντως ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Και ο λόγος είναι ότι τα κείμενά μας, η δικιά μας πρακτική, είναι να μην δημοσιεύουμε τα κείμενα όσο το Συμβούλιο δεν έχει την ευκαιρία να τα εξετάσει. Ε, να λάβουμε υπόψη μας επίσης και τις διαφορετικές αρμοδιότητες ανάλογα με το θέμα. Και τα γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Αυτή είναι η πρακτική μας αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει τίποτα άλλο. Εννοείται ότι σημειώνουμε την ανησυχία που εκφράζεται και θα τη μεταφέρουμε, εννοείται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς, γρήγορα. Σόλτ, Σόλτ. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνετε στην πράξη κατά της Χολκίν, της Continental Λαγκετ και της Γιούνιον Φενόζα που έχουν ε, παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό, έχουν διαπράξει παραβίαση και αυτό έχει καταγραφεί από την Έκοριλ, την συμβουλευτική που έχει κάνει την βιώσιμη μελέτη αντικτύπου πριν την ε, ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας. Τι κάνετε ε, επί του πρακτέου, Ματίας. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι ένα θέμα που, όπως είπα, είναι πολύ δύσκολο να συζητηθεί στο πλαίσιο της τωρινής συμφωνίας. Είναι όμως κάτι που θα μπορούμε να το εγείρουμε πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Και η κοινωνία των πολιτών θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να εκφραστεί Όπω είπα λοιπόν, ο κόσμο δεν είναι υπέροχο, το Μεξικό δεν είναι τέλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά με τη συμφωνία αυτή ε, ανοίγουμε τι δυνατότητε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού μαζί. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό, από οριζόντια μάλιστα σκοπιά υπέρ τη συμφωνία. Είμα για να ολοκληρώσουμε. Είμα! Θε να ολοκληρώσει. Ναι, ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε όμω. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε περισσότερο ποια είναι η δυσκολία. Γιατί ένα κείμενο που είναι η Συμφωνία του Μπένος Άιρες, που έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές, δεν μπορεί να ενσωματωθεί ως παράρτημα στη Συμφωνία. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω ακόμα τι φταίει για να έχουμε τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αυτή τη συμφωνία. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά την πολιτική αυτή βούληση τη ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι άλλο χρειάζεται ώστε οι ευρωβουλευτέ να έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώ διαπραγματεύεστε για κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρχει μια συνολική συμφωνία με το Μεξικό και να έχουμε στοιχεία μόνο για το εμπορικό σκέλος και όχι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα. Ας πούμε, πολλές από τις αμφιβολίες που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπήρχαν αν είχαμε όλο το κείμενο και θα μπορούσαμε και εμείς να υποβάλουμε προτάσεις πιο συγκεκριμένες για το πώς θα θέλαμε να έχει η συμφωνία. Σας παρακαλώ λοιπόν μπείτε περισσότερο σε βάθος τις απαντήσεις σας. Και κάτι ακόμα συγκεκριμένο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το κεφάλαιο αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνει η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό δηλαδή. Λοιπόν, πάλι εσείς. Thank you, Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι ερωτήσει, αλλά δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με όσα είπα προηγουμένω. Να τα πω ίσω λίγο σαφέστερα ω προ την ε, έκδοση του κειμένου, τη δημοσίευση του κειμένου δεν επικεντρώνεται μόνο στο Μεξικό. Δεν αφορά μόνο αυτή τη συμφωνία απομονωμένα, αλλά και άλλες χώρες. Είναι μια γενικότερη πρακτική και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Α πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρε αρμοδιότητε για, τα για τα εμπορικά ζητήματα. Για τα πολιτικά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στο Συμβούλιο δημιουργούνται διαφορετικές ε, ισορροπίες και άλλα μέτωπα ανάλογα με τα συμφέροντα των μεν και των δε. Η κατάσταση λοιπόν είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν αυτό δικαιολογεί το τι συμβαίνει στην πράξη, αλλά έτσι εξηγείται η σημερινή κατάσταση. Όπως είπα, σημειώνουμε τις ανησυχίες σας και θα φροντίσουμε να μεταφερθούν στους αρμοδίους Έχουμε και περιορισμούς και παρόλα αυτά έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου, να ερχόμαστε και να σας ενημερώνουμε και εσάς και την μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση και άλλους σχηματισμούς τους οποίους συνεδριάζει, υπό τους οποίους συνεδριάζει το Κοινοβούλιο. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς απλώς να δίνουμε τα ίδια τα έγγραφα, τα οποία όμως βρίσκονται στη διάθεση του Κοινοβουλίου με του ισχύοντε κανόνες μπορείτε να έρθετε και να τα συμβουλευτείτε να πάσα στιγμή. Νομίζω σημειώνουμε, σημειώνουμε τις προτάσεις σας να υπάρξει αναφορά στα ζητήματα του φίλου. Έχουμε προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσει και νομίζω ότι το τωρινό κείμενο, και καταλαβαίνω ότι δεν τα έχετε διαβάσει κιόλας, αλλά το τωρινό κείμενο τα λαμβάνει υπόψη ε, πλήρως. Ίσως ε, ίσως απλώς να μην κάνει και ρητήμνια στην διάσταση του φύλου, αλλά σίγουρα τα λαμβάνει υπόψη. Ναι. Οπότε ολοκληρώνουμε και το σημείο 25 και περνάμε τώρα στο 26. Μερκοσούρ. Όλο Λατινική Αμερική σήμερα. Νομίζω ο Ματίας Γιώργενσεν θα μας ενημερώσει και για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Παρακαλώ. Ίσως να είναι και ο κλόνος μου. Δεν είμαι βέβαιος. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Ε, πριν από δύο ρίτσες μόλις είπαμε αντίο στους ομολόγους μας από τη Μερκοσούρ. Ήταν μαζί μας όλη την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι και το Σαββατοκύριακο είχαμε διαπραγματεύσει και συνομιλίε και αυτές τις δύο μέρες, χθε και σήμερα, εντατικά όλα αυτά το τελευταίο δεκαήμερο. Καλύψαμε ένα φάσμα θεμάτων, αγαθά, υπηρεσίες, κανόνες προέλευσης, IPR, TDI, δημόσιες προμήθειες, συνοπνευματόδη, τύρι και κρασί, επιχειρήσεις, ε, αρχή της προφύλαξης και ούτω καθεξής. Είχαμε ουσιαστικές διεξοδικές διαπραγματεύσεις σε πολλούς τομείς και σε επίπεδο προϊσταμένων και σε επίπεδο τεχνικών ομάδων και τεχνικών εμπειρογνωμών. Ήταν σαφές και από τις δύο πλευρές ότι υπήρχε πολύ καλή προετοιμασία, όλοι ξέραμε, τα θέματά μας καλά και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Είχαμε πρόοδο λοιπόν στα θέματα με τη Μερκοσούρ, σε κάποια τουλάχιστον σημεία, αλλού λιγότερο. Πολύ σύντομα θα λάβετε έκθεση από την όλη συνάντηση, θα δημοσιευτεί η έκθεση όπως σε κάθε γύρο δημοτεύσεων ελπίζουμε γρήγορα και απλώς μία πρόγευση το τι σας περιμένει. Όταν λέω πρόοδο, πρόοδο είχαμε σε διάφορους τομείς, όπως τους κανόνες προέλευσης. Στα κείμενα προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε την ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη, τη διαφάνεια. Ολοκληρώθηκε αυτό το κεφάλαιο, πήγε και γρήγορα μάλιστα, σημαντικό ήταν. Μια πρόταση που εκκρεμούσε εδώ και κάποιο καιρό. Η Μερκοσούρ δεσμεύτηκε σε αυτό το γύρο ότι το κλείνουμε το θέμα. Οι δημόσιες προμήθειες, ένα θέμα που Πολλά ακόμη παρέμεναν αναπάντητα. Προχωρήσαμε, προοδεύσαμε για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λύσαμε όλα τα ζητήματα, εκτός από το θέμα της αρχής της προφύλαξης. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει συγκεκριμένη μνήμα στη δυνατότητα ενός συμβαλόμενου μέρους να εφαρμόσει 100% αυτή την αρχή. Πρέπει όμως να τα συζητήσουμε λίγο ακόμα με το, με, για να βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση. Ολοκληρώσαμε το κείμενο για την αντιμετώπιση της απάτης, σε πρόοδος πετεύθηκε στις επιδοτήσεις και επίσης το παράρτημα για τα αυτοκίνητα και το TBT. το τομείς που δεν υπήρχε τόσο πολύ πρόοδος, αλλά από τη δική μας πλευρά οι συνομιλίες πήγαν πήραν, προχώρησαν επικοδομητικά και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε στην επόμενη συνάντηση είναι επί παραδείγματι. Οι κρατικές επιχειρήσεις, οι εξαγωγικοί δασμοί και τα TBT Μετά ε, ε, υπάρχει και το κείμενο για τις υπηρεσίες που πρέπει να προχωρήσει. Υπήρχε μια σειρά από παρά τις εντατικές συζητήσεις μας να μην, εκεί δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και να έχουμε σημαντική πρόοδο. Τα τέσσερα μείζωνα ζητήματα είναι αυτά που μέχρι τώρα θα τα έχετε μάθει και απ' έξω. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις είχαμε κάποια πρόοδο Αλλά έχουμε κάποια βασικά ζητήματα για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια βασική προστασία για τα ονόματα που μας ενδιαφέρουν στη συμφωνία. Δεν μπορέσαμε όμως να έχουμε χειροπιαστή πρόοδο. Και δεν επιλύσαμε συγκεκριμένε διαφορές για κάποιε από τις γεωγραφικές ενδείξεις που θέλουμε να προστατεύσουμε. Επίσης δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε κάποια από τα θέματα πρόσβασης στην αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για τα καλακτοκομικά, τα κρασιά, το ελαιόλαδο, τα ροδάκινα. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί με βασανιστικό τρόπο και προσπαθούμε να το λύσουμε με το Μερκοσούρ είναι η υπηρεσία είναι ε, ε, το θέμα των ε, υπηρεσιών αυτών και των αυτοκινήτων, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ακόμη δεν έχουμε ε, επιλύσει το θέμα των κανόνων προέλευσης εδώ και για τα οχήματα και για τα ανταλλακτικά οχήματα. Και μετά υπάρχουν και άλλε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτέ τι δημοτεύσει. Ξέρετε ότι έχουμε πολλέ. Τα κλωστοφυντολογικά, ε, τα υποδήματα. Δεν έχουμε προχωρήσει. Υπήρξε λοιπόν αξιοσημείωτη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, αλλά έχουμε ακόμα σοβαρές ε, διαφορέ που πρέπει να κυβερνηθούν. Επόμενα βήματα. Θα δούμε. Εάν είστε τόσο εθισμένοι στο Twitter όσο και εγώ, θα δείτε τι Twitter η Επίτροπος Μάστρομ πριν από λίγο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουρουγουάης, ο κύριος Χουά, συναντήθηκε με την κυρία Μάστρομ και είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Εκεί μπορείτε να δείτε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ως προς τις συνομιλίες και τις ε, συναντήσεις. Να είστε βέβαιοι ότι παραμένουμε ταγμένοι στο σκοπό ότι αυτό από την πλευρά της Επιτροπής. Θέλουμε να πετύχουμε ε, καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία θέλουμε να έχουμε φιλόδοξη και σφαιρική και σωστά εξισορροπημένη συμφωνία στο δυνατόν γρηγορότερα. Μόλις πετύχουμε το σωστό σημείο ισορροπίας και ελπίζουμε έτσι να πείσουμε και τα κρατημέλη και το Κοινοβούλιο και τους εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και το θέμα της συμφωνίας σύνδεσης. Ναι. Μιλάμε για μια συμφωνία σύνδεσης η οποία περιλαμβάνει το εμπόριο, περιλαμβάνει και τα πολιτικά θέματα. Ε, εμείς την τελευταία συνάντηση την είχαμε τον Ιούνιο, δεν είχαμε κάποια έκτοτε. Υπάρχουν κάποια θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Ε, περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στον τομέα του εμπορίου για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε βεβαίως τη Μερκοσούρ ως οργάνωση. Είναι τεχνικά όμως αυτά τα θέματα, αλλά ελπίζουμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Κύριε Σαλαφράγκα. Ο Σε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα το λόγο και στην προηγούμενη συζήτηση, ακριβώς για να συμφωνήσω με αυτό που ζήτησε η συγκήτρια για τη συμφωνία με το Μεξικό. Εγώ είμαι υπεύθυνο από την ΑΦΕΤ γιατί ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ ανέλαβε τη δέσμευση στη συζήτηση για την κατάσταση πραγμάτων ε, στην Ένωση όταν είπε ότι θα συμμετέχει πλήρως στις εμπορικές συμφωνίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, Πρόεδρε, καταλαβαίνετε, δεδομένου αυτού η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, και εδώ να θυμίσω τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής, τη συζήτηση για την κατάσταση πραγμάτων στην Ένωση φέτος και πέρυσι, τα συμπεράσματα μετά από δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια για το ότι πρέπει η συμφωνία αυτή να καταλήξει όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα διάφορα ψηφίσματα επίσης να επιθυμίσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσαν να προχωρήσει γρήγορα αυτή η διαπραγμάτευση. Γυρνάμε γύρω-γύρω, χάνουμε χρόνο από το Δεκέμβριο πέρυσι στην ε, Υπουργική του ΠΟΕ στο Μπένος Άιρες μέχρι τώρα Έχουμε περιοριστεί σε 4-5 θέματα. Σήμερα άκουσα από τον κύριο Γιόγκενσεν ότι στον τελευταίο γύρο την προηγούμενη εβδομάδα κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί. Όμως είναι κρίμα και το λέω πρόεδρε ότι η υπουργική συνάντηση που συγκαλέστηκε τελικά δεν έλαβε χώρα. Γιατί δεν καλύπτονταν οι προϋποθέσεις Υπογραμμίζω λοιπόν ότι ο Προεδρεύων, ο Υπουργός δηλαδή της Ουρουάης που ήρθε και στις Βρυξέλλες και συναντήθηκε με την Επίτροπο, έχει κάθε καλή διάθεση. Και είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Συστήνω λοιπόν στις διάφορες πλευρές να ανασκουμποθούν, να καλυφθούν οι διαφορές σε διάφορα θέματα όπου παραμένουν και να συγκληθεί υπουργική συνάντηση πριν τα τέλη της χρονιάς, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε τη διαπραγματεύση αυτή. Και ιδιαίτερα κάνω έκκληση προς τον Επίτροπο τον κύριο Χόγκαν. Για να επιτευχθεί μια ισορροπημένη και φιλόδοξη συμφωνία, όπως είπαμε πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία από την οποία έχουν αποφελουθούν οι πολίτες μας, οι επιχειρήσεις μας και να σέβεται βέβαια απόλυτα τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε από το 2004 που είπαμε ότι θα βελτιώσουμε την προσφορά από τις δύο πλευρές. Η ελευθέρωση πρέπει να γίνει σε επίπεδα παραπάνω από το 90%. Αλλιώς θα καταλήξουμε σε ιστορική αποτυχία και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες που θα έχουμε από τον Ιανουάριο και μετά και για τις δύο πλευρές θα διευκολύνουν μια επιτυχή έκβαση μια διαδικασία που έχει κρατήσει τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν έκκληση κάνω προ την Επίτροπο Μάριστρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουν γρήγορα, να διαλυθούν τα τεχνικά προβλήματα και να συγκληθεί η Υπουργική Συνεδρίαση μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έχει αναφερθεί στην Επιτροπή μας και προηγουμένως, τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες μιας τεράστιας ευκαιρίας που έχουμε και οδεύουμε προς την επίταξη της συμφωνίας αυτής. Ω πρόεδρο λοιπόν τη αντιπροσωπεία στι ε, τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βραζιλία, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη σημασία τη συμφωνία αυτή για μια χώρα με τι διαστάσει τη Βραζιλία. Γι' αυτό υπήρχε και στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βραζιλία από το 2007, ε, τόσο σημαντική που η Βραζιλία δεν είναι απλώς σημαντική στον κόσμο λόγω κόσμου, αλλά και πληθυσμού και παραγωγής και είναι και η μεγαλύτερη οικονομία της Μερκοσούρ. Γι' αυτό η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας είναι σημαντική και γενικότερα είναι σημαντική η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούλ. Είναι σημαντικό αυτή η σφαιρική συμφωνία να επιτευχθεί γρήγορα διότι η νοτιοαμερικανική αγορά πρέπει να ε, είναι μια αγορά που έχουμε πρόσβαση χωρίς τάσεις προστατευτισμού και να προαχθούν οι σχέσεις της Ευρώπης με την Λατινική Αμερική και την Βραζιλία πιο συγκεκριμένα. Έχουμε όμως και κάποιους ενδιασμούς να εκφράσω κυρίως για όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία, την έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων με τη νέα κυβέρνηση να αναλαμβάνει και να μην προωθεί αρκετά την Μαρκοσούρ. είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες για το τι θα συμβεί ε, στις σχέσεις μας στην επόμενη φάση μεταξύ των δύο αυτών γεωγραφικών περιοχών. Επίσης, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο Ομοσπενδιακός Υπουργός Οικονομικών ε, της Βραζιλίας στην επόμενη φάση και είπε ότι ε, ο υπουργό δεν θα εκφράζει τις ίδιες επιθυμίες με την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί θυμάμαι μια συνέντευξη του ε, Προέδρου Μπολσονάρα από τις 5 Οκτωβρίου που έλεγε ότι οι εμπορικές σχέσεις με τις υπόλοιπες ε, περιοχές του κόσμου θα πρέπει να γίνουν με κεντρικό τρόπο και είπε ότι οι αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής της χώρας θα εξαρτηθούν και από τις συζητήσει και τις ε, ισορροπίες ε, ε, της μελλοντική κυβέρνησης και το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν κάποια επισιοδοξία, όμω οι πρωταγωνιστέ τη πολιτική ζωή ε, από την άλλη πλευρά του ωκεανού δεν θα είναι πια οι ίδιοι. Θα τα δούμε λοιπόν μάλλον καλύτερα του χρόνου ε, που θα έχουμε και τι ευρωεκλογέ. Ελπίζω, ολοκληρώνοντα, ότι οι νέοι πρωταγωνιστέ δεν θα πάψουν να εργάζονται υπέρ τη ε, επίτευξη αυτή τη συμφωνία διότι αυτό μου φαίνεται ότι είναι το πλέον επίγον και σημαντικό και για τις δύο περιοχές του κόσμου αυτούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδης, ο κύριος Ντάντι για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, πήγαμε σε επίσκεψη με την αντιπροσωπεία της Μερκοσούρ στην Παραγουάη και Ουρουγουάη και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικά προβλήματα πολύ σοβαρά. Διότι πέραν των ωραίων κουβεντών που, και λόγων που όλοι λέμε, μιλάμε για δύο χώρες που ουσιαστικά δεν τη θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ας πούμε, ας είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν έχει επιτευχθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία και σήμερα δεν είμαστε σε θέση να έχουμε πραγματικά βήματα πρόοδου από τι συμφωνίε αυτέ, το είπε και ο κύριο Γιώργενσεν. Δεν μπορούμε να θεωρούμε πρόοδο αυτά που έγιναν ε, ε μέχρι τώρα. Από τα πέντε προβλήματα μα έχουν μείνει τα τέσσερα. Δηλαδή, πέρασαν δέκα μέρε για να λύσουμε μισό πρόβλημα. Τα σημαντικά που είναι οι γεωγραφικέ ενδείξει, οι θαλάσσιε υπηρεσίε, το κρασί, το ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά κυρίω. Αυτά ούτε που τα κομπήσαμε. Τα αυτοκίνητα ούτε καν. Ε, ίδιες και παράλλαχτα μείναν οι θέσει τη Μερκοσούρ. Πού είναι λοιπόν η πρόοδο ε, με τι δημόσιε προμήθειε. Εντάξει, σημαντικό είναι και αυτό, αλλά για το χρόνο που έχουμε αφιερώσει, διότι έχουμε να κάνουμε με προθεσμίε εδώ που πιέζουν ε, και το Ευρωκοινοβούλιο έχει και ευρωεκλογέ όπου να είναι. Αλλά μόλι ανέλαβε και η νέα κυβέρνηση στην μεγαλύτερη χώρα, τη Βραζιλία. Άρα δεν σημαίνει ότι οι θέσει τη χώρα δεν θα αλλάξουν σε τίποτα, ούτε ότι δεν θα επηρεαστούν ε, οι θέσει των υπόλοιπων χωρών τη Μερκοσούρ. Α είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, εντάξει, αλλά η αισιοδοξία ε, σταματάει πια και στερεύει μπροστά στην τελευταία κλειστή πόρτα. Εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο κάθε προσπάθεια που μπορούσαμε την κάναμε. Όμω πρέπει να ε, σημειώσουμε ότι παρά την αφοσίωσή μα, τα βήματα προόδου, για τα προβλήματα αυτά δεν βρήκαμε εγώ δεν βρήκα σε καμία από τις χώρες αυτές καμία ανταπόκριση. Ας πούμε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το λέω ως παράδειγμα, αλλά για τα θέματα αυτά, ξέρω εγώ, η σαμπάνια της Ουρουγουάης και το παρμιτζάνο ρετζάνο, παρμεζάνα της Ουρουγουάης, πώς θα αλλάξουν όνομα. Είναι πολύ δύσκολα θέματα αυτά, αν δεν υπάρξει διάθεση υποχώρησης από κάποιον ή μια διάθεση συμβασμού. Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν. Ε, ας συνεχίσουμε, ας προσπαθήσουμε κι άλλο, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι και η πολιτική βούληση που υπάρχει εδώ. Ε, ένα βήμα πρόοδου το κάναμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. από τα θέματα που είχαμε εντοπίσει πριν από 10 μήνες όμως ως ζωτική σημασία, έχουμε μείνει στο ίδιο σημείο. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον κύριο Γιώργενσεν είναι ξέρει ποια θα είναι η θέση της Βραζιλίας. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Αλλά πριν προχωρήσουμε, αυτέ οι διαπραγματεύσει που φαίνεται ότι θα ολοκληρώνονταν πριν από εδώ και 10 μήνε, μείναν στο ίδιο επίπεδο. 10 μήνε μετά. Ευχαριστούμε κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Όμως μετά τη χθεσινή συζήτηση εδώ στην ημερίδα για το εμπόριο πρέπει να ε, προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό σε μεγαλύτερο βάθος. Συζητήσαμε για τη διοντολογία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούμε ξαφνικά να υποκριθούμε ότι θα συνεχίσουμε business as usual με την νέα βραζιλιανική ε, κυβέρνηση. Ε, όταν τίθενται σε κίνδυνο ζητήματα όπως είναι η βιωσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε την αποψήλωση των δασών του ε, Αμαζονίου για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η καλλιέργεια σόγιας και άλλων φυτών. Αυτά δεν μπορεί να είναι θέματα τα οποία θα μπορούσαν να αγνοηθούν στην διαπραγμάτευση. Όλα αυτά που είπατε σωστά είναι ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια και δυσκολία θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ναι, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συνολική εικόνα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο της Μερκοσούρα αλλά και του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Είπαμε και, στο, και στην περίπτωση του Μεξικού ότι ιδανικό κόσμος δεν υπάρχει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιτρέψουμε την επιδείνωση αυτού του μη ιδανικού κόσμου και να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θυμάμαι ε, ότι με τον κύριο Σαλαφράγκα ως εισηγητή τότε είχαμε βρεθεί, με την, ε, είχαμε βρεθεί στην Αργεντινή και εκεί είχαμε ήδη καταλήξει το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα, να σημειωθεί συγκεκριμένη προόδος ε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν δεν έχει υπάρξει σημείο, πρόοδος. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι με τις νέες ηγεσίε ε, στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής μπορούμε να σημειώσουμε αυτή την πρόοδο που δεν επετέχει τα δύο τελευταία χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες να συνεχιστούν αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση να ξεκαθαρίζεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτουμε για τη σύναψη ε, εμπορικών συμφωνιών. Κύριε Μινέρ, ευχαριστώ. Σήμερα μια η Ολλανδική εφημερίδα να φέρει ένα άρθρο που λέει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Γιατί τελικά θέλουν ε, να κάνουν εξαγωγές από τη Μερκοσούρ προϊόντων που θα καταστρέψουν τους μικρούς παραγωγούς και επίσης και για όλα αυτά για τα δάση και για τον πρόεδρο τον καινούργιο της Βραζιλίας ο οποίος καταστρέφει τον Αμαζόνιο τα δάση του Αμαζονίου που θα εξαφανιστούν. Είναι επίσης, γίνονται φοβερές παραβάσεις και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της βιοπικιλότητας. Το δάσος του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο σε ολόκληρη τη γη και δεν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα κατά 1,3 γίγατον το χρόνο θα αυξηθούν οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα αν καταστραφεί το δάσος αυτό. Λοιπόν, μια τέτοια, με μια τέτοια προσωπικότητα όπως είναι ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας δεν πρέπει να έχει δουλειές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Είμα. Έχω μια ερώτηση, παρακαλώ. Πώς εκτιμάμε την Προεδρία του κύριου Μποσενάρο στην διαδικασία διαπραγματεύσεων της συμφωνίας με τη Μερκοσούρ. Όπως συμβαίνει με πολλές του δηλώσεις, ο πρόεδρος ποσενάρο φαίνεται ότι ακολουθεί την πολιτική Τραμπ. Είδαμε πώς έκανε διαπραγματεύσεις για την ναύτα ο Τραμπ. Έκανε δύο διμερείς συμφωνίες αντί για μία περιφερειακή. Μπορεί να κάνει το ίδιο κι αυτός μπορεί να έχει μία στρατηγική αντί για μία περιφερειακή συμφωνία όπως θέλουμε εμείς και που θα ήταν πολύ θετικό για τη Μερκοσούρ και για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική αλλά και την Ευρώπη. Μήπως θα προσπαθήσει να επιβάλλει τη δικιά του οικονομική κυριαρχία κάνοντας διμερείς συμφωνίες με τις διάφορες πλευρές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η κυρία Ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρους της Δίτα Σαράντσοβα, που είναι σκιώδης συγκήτρια. Η Δίτα λοιπόν επαναλαμβάνει την άποψή τη, που είναι και άποψη τη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι στηρίζουμε την κατάληξη τη εμπορική αυτή συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χαίρεται γι' αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που δεν έχει κλείσει. Παρόλα αυτά, ανησυχεί ε, για το γεγονός ότι συνεχίζονται και διονύζονται οι διαπραγματεύσεις. Στην αρχή ήταν η προθεσμία το 2017, μετά 2018, Μάρτιος, Ιούλιος. Η πολιτική συμφωνία πρέπει να γίνει. Μπορεί να υπάρχει συμφωνία του G20 στο Buenos δεδομένου και να μην έχουμε μη συμφωνία ενώ έρχονται οι ευρωεκλογέ για το ΚΑΡ στη Γεωργία. Πρέπει να γίνει σαφέ, τελικά αν θα προχωρήσουμε στη συμφωνία ή όχι. Και ποιε θα είναι οι επιπτώσει αν δεν υπάρχει συμφωνία ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την εμπορική μας συμφωνία με το Μεξικό Τώρα θέλουμε να εξυγχρονίσουμε και την εμπορική συμφωνία με τη Χιλή. Συμφωνίες από τις οποίες τα ωφέλη είναι πολλά και για τις λογοπεριοχές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ όμως δεν φαίνεται να καταλήγουμε. Ελπίζει την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα γιορτάσουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την νέα συμφωνία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής όλες οι συμφωνίες που συζητήσαμε που είναι όλες πολύ φιλόδοξες πρέπει να ολοκληρωθούν και να συναυτούν πριν από τις ευρωεκλογέ. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ε, που επικρατεί στη Βραζιλία για τους γεωργούς. Σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν θεωρώ ότι θα τους βοηθήσει. Λαμβανωμένη υπόψη και της πολιτικής κατάστασης που πλέον επικρατεί στη χώρα. Κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το συζητήσαμε και στην περίπτωση του Μεξικού. Τα ίδια ισχύουν και με τις χώρες Μερκοσούρ ποια ακριβώς θα είναι η αντίδραση από πλευράς μας όταν θα διαπιστώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μιας και αναφέρατε σε, τόσ, σε τόσες πολλές προόδους που έχετε κάνει, βιωσιμότητα, πείτε μας κάποια πρακτικά παραδείγματα που επιτύχατε. Τι τελικά τόσο ρηξικέλευθο συνέβη σε αυτούς τους τελευταίους γύρους διαπραγμάτευσης για να μας πείτε και να μας λέτε ότι πραγματικά σημειώσατε πολύ μεγάλη ε, πρόοδο. Merci. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, ή που Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πληροφορίες που εμείς δεν διαθέτουμε, γιατί ξέρουν ότι ο νέος πρόεδρος που εξελέγει στη Βραζιλία δεν θα αναλάβει καθήκοντα την ημερομηνία που κανονικά πρέπει να αναλάβει καθήκοντα, οπότε τότε ακόμα κι αν έχω διάφορες επικρίσεις για τη Μερκοσούρ, κυρίως για τη Γεωργία, για το περιβάλλον, αλλά ε, τότε υπάρχει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μπολσονάρο δεν θα είναι ποτέ πρόεδρος. Αν όμως δεν είναι έτσι, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορεί να μας λένε ότι όταν έχουμε δημοκρατία διαπραγματευόμαστε, όταν δεν έχουμε δημοκρατία κινδυνεύει η δημοκρατία, πρέπει να διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή πάντα πρέπει να διαπραγματευόμαστε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών, γιατί ελεύθερε συναλλαγέ είναι η λύση τόσο για τι αυταρχικέ κυβερνήσει όσο και για τι δημοκρατικέ. Ε, όχι, δεν γίνεται. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται απέναντι σε δυσκολίες μετά τη Συμφωνία των Παρισίων ε, δεδομένη της αποψήλωση των δασών, ε, των προβλημάτων στη Γεωργία. Και εδώ είμαστε έτοιμοι να ε, καταλήξουμε σε συμφωνία με κάποιον ο οποίος δημόσια ανακοίνωσε ότι θα αφήσει να καταστραφεί ο Αμαζόνιος και ότι θα επιτρέψει σε όποια χώρα θέλει να πάει να φτιάξει, ε, να παράγει, να καλλιεργήσει τέλο πάντων σόγια εκεί πέρα, θα μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Μα τι είναι αυτά. Εμείς πρέπει να πούμε ότι δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία με ηγέτη ο οποίος δεν δέχεται τη συμφωνία των Παρισίων. Μα κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε σε μια τόσο σημαντική στιγμή πολιτικά τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο για τη Λατινική Αμερική. Αν δεν σταματήσουμε διαπραγματεύσεις, δεν παγώσουμε τις διαπραγματεύσεις για να δούμε ποιο είναι τελικά το πλαίσιο αρχών και αξιών βάσει των οποίων καταλήγουμε σε εμπορικέ συμφωνίε, τότε δεν καταλαβαίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλήθεια, όπω είπα πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάποιε πληροφορίε για τον νέο Βαρζιλιάνο πρόεδρο που εμεί να μην διαθέτουμε. Τελευταίος, ο κύριος Ντάτμαθ. Ευχαριστώ. Τι να σας πω είναι θέμα αρχής, όπως καταλαβαίνετε. Ε, εν πάση περιπτώσει, έχω κάποιες ερωτήσεις. Και λυπάμαι από μου ο τελευταίος, γιατί θα ήθελα απαντήσεις. Ο κύριος Αντώ είπε ότι ο Μπαλσονάρο ο εκλεγμένο. το είπε. Και ίσως δεν του αρέσει. Εντάξει, μπορώ να συμφωνώ κι εγώ μαζί του, αλλά ο Μπολσανάρο δεν έχει αναλάβει ακόμα καθήκοντα. Είναι ακόμα στις υποσχέσεις. Και ξέρουμε τι γίνεται με τους εκλεγμένου, Βέβαια πάντα εξαιρούνται οι παρόντε, αλλά οι προεκλογικέ υποσχέσεις δεν σημαίνουν και πολλά μετά. Οπότε τώρα έχουμε το νέο δόγμα Ζαντό, ότι βάσει των υποσχέσεων να παίρνουμε αποφάσεις. Δεν ξέρω, να το συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί. Και στην ίδια γραμμή με την κυρία Μινέρ, λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε business με τον πρόεδρο Μπολσενάρο, τον εκλεγμένο προσθέτω εγώ. Ε. Οπότε όμως τίθονται τα ερωτήματα, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Με αυτά τα κριτήρια τελικά με ποιον κάνετε business και με ποιον δεν κάνετε business. Καταλαβαίνετε ότι ο κατάλογος ε, κινδυνεύει να είναι πάρα πολύ μικρός τελικά. Εδώ έχουμε ε, εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Με κάθε σεβασμό, εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από τη στάση του ΕΛΚ όσον αφορά την στάση του στο καταλωνικό ζήτημα που βάλαν στη φυλακή τους πολιτικούς. Δεν ξέρω θα ήθελα κάποια διαφώτιση από τους συναδέρφους. Ε, αν όχι σήμερα, κάποια άλλη στιγμή. Πολύ θα ήθελα να μου απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Φίσας. Θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο ότι δεν βάζουμε στη φυλακή κανένα καταλανό ε, αποσχιστή. Η πολιτική που είναι στη φυλακή δεν είναι ε, πολιτικοί κρατούμενοι, είναι πολιτικοί που βρίσκονται στη φυλακή γιατί παραβίασαν το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, λέει ο Πρόεδρο. Τώρα, ο πρέσβη τη Ουρουάη, που εκπροσωπεί τις χώρες Μερκοσούρ εδώ σήμερα. Για ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας Διεθνούς Εμπορίου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ πολύ και τον Ματίας και τον Αντριάνου για τις παρεμβάσεις τους. Επιβεβαιώνω ότι στις 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες είχαμε εντατικές ημερίδες εργασίας με τους επικεφαλείς των διαπραγματεύσεων και τις τεχνικές ομάδες της Μερκοσούρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να ξεμπλοκάρουμε πια τα διάφορα θέματα στα οποία είχαμε κολλήσει και που ήταν τεχνικής φύσης. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιζόταν από μια υπουργική συνάντηση με τις Επιτρόπους Μάλστρομ και Χόγαν, εδώ στις Βρυξέλλες ε, πάντα, για να συζητηθούν τα πέντε πιο ευαίσθητα ζητήματα και να δούμε πώς μπορούσαμε να τα χειριστούμε πολιτικά. Αν πετύχαινε αυτή η συνάντηση, θα ολοκληρωνόταν και αυτή η μακρά διαπραγματευτική διαδικασία. Όντως, λοιπόν έγινε πρόοδος σε πολλούς τομείς και έκλεισαν κάποια σημαντικά ζητήματα. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν από τον Ματίας. Όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι τα θέματα αυτά που έκλεισαν ήταν κυρίως ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στην ευελιξία της Μερκοσούρ. Παραμένουν διαφορές όμως σε κάποια άλλα ζητήματα που θεωρούνται τεχνικά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση την πέμπτη το απόγευμα ε, σταμάτησε την ε, συνάντηση αυτή. Έτσι έγινε πίεση προς τους διαπραγματευτές να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε σύγκληση. Η παρουσία των Υπουργών θα βοηθούσε να πάρουμε την πολιτική κατεύθυνση προκειμένου να έχουμε λύση. Ο Νίνο Μπόα, Υπουργό Εξωτερικών και προσωρινά πρόεδρος της Μερκοσούρ, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμό Αυτό ήθελαν οι χώρες Μερκοσούρ. Και μίλησε με την Επίτροπο Μάλστρομ και τη Σάντρα Καλίνα που ήταν ε, διαπραγματευτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικά αποτελέσματα και οι δύο πλευρές είπαν ότι θέλουν να συνεχιστεί η διαδικασία σε τεχνικό επίπεδο και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες και ρεαλιστικές λύσεις ώστε να συγκληθεί η Υπουργική Συνάντηση πριν από τα τέλη της χρονιάς για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαπραγμάτευση αυτή. Τώρα που μιλάμε, προσπαθούμε να βρούμε ημερομηνίε το Δεκέμβριο και ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε. Θεωρούμε ότι είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Αλλιώς ποιος ξέρει πώς και πότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, υπογραμμίζοντας ότι τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Ματίας, όπου δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος τη βδομάδα εκείνη, είναι γεωγραφικές ενδείξεις, θαλάσσιες υπηρεσίες, χαλακτοκομικά και θέματα που έχουν να κάνουν με ποσοστώσεις γεωργικών προϊόντων που ενδιαφέρουν τη Μερκοσούρ. Γι' αυτά πρέπει να πούμε ότι εντοπίστηκαν αυτά τα θέματα από τους υπουργούς ώστε να ε, τύχουν ε, εξέτασης από τους ίδιους τους υπουργούς. η τεχνική δηλαδή παρά τις μεγάλες ε, προσπάθειες που έκαναν έφτασαν στα όρια τους για αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Αντριάνου για αυτά που είπε και συμφωνώ μαζί του για την εκτίμησή του. Οι χώρε Μερκοσούρ είμαστε διατεθειμένε να καθίσουμε ανα πάσα στιγμή ώστε να ολοκληρωθεί μια για πάντα η συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πρέπει έχει κάποιε ερωτησούλε να απαντήσει. Ματίας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και Ίσως, ξεκινώντας από το τέλος, μετά από όσα είπε ο φίλος μου, ο πρεσβευτής από την Ουρουάη. Δεν υπάρχει θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέκοψε υπουργική σύνοδο από την πλευρά της Επιτροπής. Αναφέραμε την προθυμία μας και τη διατηρούμε να έχουμε υπουργική σύνοδο όταν υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε κάπως περιορίσει τα προβλήματα που παραμένουν αναπάντητα και να είναι όριμα τα πράγματα και κατάλληλα για μια υπουργική σύνοδο. Η κατάσταση ακόμα δεν είναι τέτοια. Αυτό αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην αλληλογραφία μας και τις ανταλλαγές μας με τους υπουργούς. Μια υπουργική θα μπορούσε να οργανωθεί μόνο αν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει, παρόλο, και το αναγνωρίζω αυτό, που έγιναν σοβαρές προσπάθειες και από την πλευρά της Μερκοσούρ και από τη δική μας. Τώρα, για κάποια από τα σχόλια σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ήταν ε, πολύτιμη. Το Ευρωκοινοβούλιο βοήθησε στο να βρούμε τον κατάλληλο ρυθμό για να προχωρήσουν οι και να μπορέσουμε να οδεύσουμε προς ολοκλήρωση. Τη χρειαζόμαστε την υποστήριξη, γιατί θα πρέπει να λάβουμε σκληρές αποφάσεις, όχι μόνο για τη Μερικοσούρ και για να λάβουμε υπόψη και τις ευαισθησίες της άλλης πλευράς και να τους δώσουμε και κάτι, κάτι που να αξίζει και για αυτούς. Να μην ξεχνάμε ότι και αυτό πρέπει να συμβεί. Ολοκλήρωση. Ωραία, ναι. Να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν συντομότερα. Πώς να ολοκληρώσουμε όμως όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά ζήματα, ζητήματα όπω η αρχή της προφύλαξης που δεν έχει επιληθεί και εκεί που έχουμε ζητήσει ουσιαστικά για την, ε, από τη Μερκοσούρ να λάβει υπόψη την σημαντικότητα αυτή για, αρχή για μας και για τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις εμβληματικότερες για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τις έχουμε καλύψει, δεν έχουμε εγγύησει από το Μερκοσούρ, ούτε ικανοποιητικέ λύσεις για το πώς θα προστατεύονται. Και για τους κανόνες προέλευσης που προτείνει η Μερκοσούρ για την αυτοκινητοβιομηχανία, με αυτά που προτείνονται, το εμπόριο γίνεται σχεδόν αδύνατο. Είναι πολλά λοιπόν τα περίπλοκα ζητήματα που ακόμη έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για την βιώσιμη ανάπτυξη, τι εκλογέ στη Βραζιλία και το τι θα γίνει. Ναι. Είναι θέμα το τι θα γίνει με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Μπολσονάρου στη Βραζιλία και το τι κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Όμω το θέμα είναι τι κατεύθυνση θέλουμε να δώσουμε και εμεί τα πράγματα. Θέλουμε να κλειδώσουμε και να μπλοκάρουμε την ε, Βραζιλία ξεχνώντας τις ε, οικειοθελείς ε, πολυμερείς συμφωνίες ή θα προσπαθήσουμε να τους παρασύρουμε σε κάτι θετικό στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων ας πούμε. Θέλουμε να αναζητήσουμε χώρους συνεργασίας μαζί τους ή όχι. Αυτό είναι καθοριστική σημασίας το κεφάλαιο εμπορικών ε, συναλλαγών με χώρες που υπογράφουν, ε, εφαρμόζουν με συνέπεια και δεν παρακλίνουν των προτύπων των συμβάσεων του ΑΕΛΟ ή των βασικών πολυμερών συμφωνιών είναι κάτι που νομίζω ότι τους πάει όλους στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά είναι πολιτική επιλογή. Δεν ξέρω τι πληροφορίε έχει το Ευρωκοινοβούλιο και δεν ξέρω αν είναι διαφορετικέ από αυτέ που έχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, εμεί αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και τώρα. για το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης και σε σχέση με όσα προτάθηκαν προηγουμένως. Σε αυτό το κεφάλαιο της συμφωνίας αυτής Έχουμε κάτι πολύ παρόμοιο με όσα είχαμε στις ε, πολύ καλές συμφωνίες μας ως τώρα. Αυτά μας ενέπνευσαν. Και αυτό που πετύχαμε αυτή τη φορά είναι να έχουμε συμφωνίες για την διοργάνωση πάνελ ή του είδους τι είδους διαδικασίες μπορούμε να εφαρμόσουμε. Αυτά. Παντός ακούω και καταγράφω τα μηνύματα του Ευρωκοινοβουλίου. Καταλαβαίνω ότι για σας είναι καταπήγον, θα φροντίσω να μεταφερθεί στους ε, προϊσταμένους. Ε, Κέσον, έχετε κάτι να προσθέσετε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την έντονη συζήτηση. Αλλά ε, θα ήθελα να συμφωνήσω κατά πολύ με όσα είπε ο συνάδελφό μου, ο Ματία, από τη Γενική Διεύθυνση Trade. Όχι τόσο πολύ για το αν θα το συμπαρασύρουμε εδώ. Μιλάμε για μια συμφωνία σύνδεση και αμοιβαίω έχουμε δεσμευτεί να λύσουμε ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά όχι μόνο για το εμπόριο το εμπόριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή, αλλά και πολιτικές δεσμεύσεις που υπάρχουν για να προστατευτεί το κάτω σε δικαίωμα δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμμετοχή σε πολιτικά, οικονομικά, ε, κοινωνικά ε, και από τι δύο πλευρέ θέλουμε αυτά να προωθηθούν. Και να μην ξεχνάμε ότι οι χώρε με τι οποίε διαπραγματευόμαστε είναι αρκετά αναπτυγμένε πλέον. Δεν είναι υποανάπτυκτε, ούτε αναπτυσσόμενε ούτε έχουν καμιά περίεργη κυβέρνηση, ακόμη και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις για την κυβέρνηση της Βραζιλίας. Αλλά μιλάμε για κοινωνίες με φορείς πολύ ισχυρού και στον οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό. Με διαφορετικές ενδεχομένως απόψεις ε, και που έχουν άποψη και μάλιστα πολύ σοβαρή για τις συμφωνίες αυτές σε σχέση με το παρελθόν. Στη συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα την αποφασίσουν οικονομικέ δυνάμει που έχουν πολύ διαφορετικέ τάσει και συμφέροντα από αυτά που νομίζουμε εμεί και έχουν διαφορετικά πράγματα να προσπιστούν στι χώρε του. Η αξία λοιπόν τη συμφωνία αυτή ε, πηγαίνει πολύ παραπέρα από το εμπόριο απλώ, τα αγαθά και τι υπηρεσίε. Είναι μια δέσμευση για ένα μοντέλο δημοκρατικό, ένα μοντέλο ανθρωπίνων αξιών. Και όχι μόνο σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την κοινότητα των πολιτών με όλο το σύστημα των χωρών αυτών. Είναι σημαντικό να βρούμε την σωστή διασύνδεσή μας, τον τρόπο να, να σχετιστούμε με τις κοινωνίες των χωρών αυτών. Τώρα για τις επιθέσεις, τις πιέσεις που δέχεται το μοντέλο αυτό, οι ίδιε δυνάμει υπάρχουν και στι χώρε αυτέ, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τι αντίστοιχε δυνάμει των δικών μα, που στι χώρε αυτέ προσπίζονται τι δικέ μα αξίε. Ωραία. Και ο κύριο Σαλαβάνκα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Έφυγε ο κύριος Στόρμου, το απάντησε βέβαια ο κύριος Φίσας όταν μίλησε για τους αποσχιστές ε, της Καταλωνίας. Βλέπετε, αντίθετα με την ε, Σκοτία, η Καταλωνία ποτέ δεν ήταν ένα ξεχωριστό ε, βασίλειο, ήταν στην Αραγωνία. Άρα είναι μια από τις αυτόνομες περιφέρειες που επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι χαίρεται από τη μεγαλύτερη αυτονομία σε ολόκληρη την Ευρώπη. πρέπει κανείς να τηρεί τον νόμο. Μόνο αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου αν δεν τηρείται ο νόμος. Αυτά για την Καταλωνία. Τώρα για το θέμα που μας απασχολεί. Είναι σημαντικό να σταθμίσουμε την πραγματικότητα, χωρίς ε, να υπερβάλλουμε αλλά και χωρίς να κρύβουμε πράγματα. Το τμήμα της συνεργασίας έχει περίπου ολοκληρωθεί και το εμπορικό πριν από την τελευταία συνάντηση είχε ολοκληρωθεί κατά 90%. Έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις στον τελευταίο γύρο. Δεν ξέρω η Κομισιόν σε τι ποσοστό θεωρεί ότι υπάρχει πρόοδος. Εγώ νομίζω ότι είναι της τάξης του 3 με 4%. Οπότε θέλω να καθησυχάσω τον κύριο Ντάντι, τον συνάδελφο, γιατί υπήρξαν σημαντικές, υπήρξε σημαντική πρόοδος και για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για την αυτοκινητοβιομηχανία και για τα ανταλλακτικά. Λίγα θέματα μένουν ακόμα. Θα έλεγα μάλιστα, ας είμαστε ειλικρινεί απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη. Είμαστε υπέρ του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας με την Κούβα. Και όπου να είναι, θα δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη και για το Βιετνάμ. Εδώ πάνω από 20 χρόνια έχουμε τέτοια συμφωνία με τη Μερκοσούρ και δεν είναι δυνατόν επειδή μια εφημερίδα σε μια χώρα μέλος έγραψε κάτι ή επειδή ακούμε ότι ξέρω εγώ τι με τις εκλογές όπως έχουμε τώρα στη Βραζιλία. Θα έλεγα στο συνάδελφο ότι ναι, συμμερίζομαι την ανησυχία του για το ότι η Βραζιλία εγκαταλείπει τη Συμφωνία των Παρισίων. Είναι ανισχυτικό. φυσικά, όπως και τα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται σε βασική ρήτρα στις συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, εγώ θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον συγγνώμη, στην Επιτροπή μας, να μην είμαστε τόσο αλαζόνες. Τις συμφωνίες δεν τις και τους όρους δεν τους κάνουμε μόνοι μας, είναι δύο πλευρές. Και δεν καθορίζεται η διαδικασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν κάποιο είναι σε διαπραγματεύσεις διμερός, πρέπει να δείξει την επιθυμία να επιτευχθεί συνένεση. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική στρατηγικά, εμπορικά, πολιτικά και οικονομικά. Υπάρχει εδώ μια ευκαιρία να καταλήξουμε πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Ζητώ λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια ώστε και δύο πλευρές πρώτον να συμφωνήσουν για την οργάνωση αυτής της Υπουργική συνάντησης και δεύτερον να μην πάμε πίσω σε σχέση με τόσο έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Υπάρχει μια χώρα που είναι στη Μερκοσούρ και που κάνει πίσω σε κάποια πράγματα να μην μας αποκλείσει αυτό από τη συμφωνία. Αλλιώς νομίζω ότι όλοι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και αυτό δεν θα είναι καλό. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε το σημείο 26 και περνάμε αμέσως στο 27 από τη Νότια Αμερική στην Βόρεια Αμερική τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ που επίσης αποτελούν σημαντικό στοιχείο του εμπορίου και των ενδιαφερόντων μας. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Επιτρόπος μας βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για να συνομιλήσει με τον ομολογό του. Θα διαβάσετε στον τύπο ότι ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησε την έκθεση για τους δασμούς στα οχήματα, την γνωστή έκθεση 232 με τους ε, συμβούλους του και συλλέξαμε και κάποιες εμπειρίες σχετικά με τις συνομιλίες μας με εκπροσώπους των ΙΠΑ οι οποίοι φαίνεται ότι προχωρούν σε αυτήν την μάλλον σκληρή στάση τον ΗΠΑ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν, ε, στάση που ήδη έχουν τηρήσει, στο χάλιβα, στο ε, αλουμίνιο, τώρα κάνουν το ίδιο στα οχήματα, προφανώς για να αποσπάσουν κάποιες υποχωρήσεις ή παραχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός μας είναι να ενημερωθούμε, για τα όσα συνέβησαν καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις που αναμένονται στο μέτωπο των εμπορικών συνομιλιών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου εδώ μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε στα τέσσερα βασικά θέματα που συζητούμε σχετικά με την εφαρμογή της κοινή δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους δύο προέδρους τον Ιούλιο έπειτα από τις συνομιλίες που είχε η Επίτροπος Μάλστρομ με τον ε, πρέσβη Λάιτχάισερ. Θέλω να στραφώ πρώτα στο ζήτημα των βιομηχανικών δασμών. Ξέρετε ότι η κοινή δήλωση δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής εμπορική διαπραγμάτευση την οποία μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή με τις ΣΥΠΑ, είναι η διαπραγμάτευση για την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε στις, Ευρω... στις Ηνωμένε Αμερικής από την αρχή ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εργασίες της ομάδας εργασίας προκειμένου να ε, διευθετήσουμε τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Οι ΙΠΑ μας είπαν ότι δεν επίγονται ιδιαιτέρως. Στη συνέχεια οι ΙΠΑ αποφάσισαν να κοινοποιήσουν προς το Κογκρέσο την επιθυμία τους να ξεκινήσουν διαβούλευση για την έναρξη διαπραγματεύσεων και ε, μας ενημέρωσαν ότι οι διαβουλεύσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη ε, και έως ότου ολοκληρωθούν δεν μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με εμάς. Για τους δασμούς αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έχω κάτι νέο να σας πω. Η Επίτροπος ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι ο μόνο είδο διαπραγμάτευση στο οποίο μπορούμε να, να μπούμε είναι, είναι μια διαπραγμάτευση που θα αφορά τους ε, βιομηχανικούς δασμούς. Ο πρέσβης τον είπα, μας είπε ότι περιμένει το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με το Κογκρέσο και η διαβούλευση αυτή θα ολοκληρωθεί όχι πριν τον Ιανουάριο. Μόλις μάθουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και, και εσάς σε σχέση με τους βιομηχανικούς δεσμούς. Το βασικό ζήτημα που μας απασχόλησε στην εκτελεστική ομάδα εργασίας είναι κανονιστικά θέματα. Προσδιορίσαμε το βαθμό στον οποίο μπορούμε να σημειώσουμε προόδο στη βάση των κοινών μας συμφερόντων και ε, μπορώ να σας πω ότι οι συζητήσεις ήταν θετικές, ε, συμμετείχαν ρυθμιστικές αρχές και των δύο πλευρών ε, πριν από την συνάντηση της Επιτρόπου με τον ε, Πρέσβη. Ε, είχαμε στην Ουάσιγκτον μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που, ε, ε, στην οποία εκπροσωπούνταν και διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίστοιχοι ομόλογοι υπήρχαν και από την πλευρά των ΙΠΑ και η ομάδα εργασίας αυτή προσδιορίσε τρεις πιθανούς τομείς όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Οι τρεις αυτοί τομείς είναι τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η κυβερνοασφάλεια. Μπορώ να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες, αν ε, επιθυμείτε να τις λάβετε. Αυτοί είναι οι τρεις τομείς που προς το παρόν έχουμε προσδιορίσει ότι πράγματι προσφέρουν ε, καλές δυνατότητες ε, προόδου, Επίση, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομεί στου οποίου έχουν ξεκινήσει απλώ οι συζητήσει, αλλά εκεί φαίνεται ότι θα χρειαστούν περισσότερε συζητήσει για να σημειωθεί η πρόοδο. Μιλάμε για την αξιολόγηση συμμόρφωση, για τα βιομηχανικά πρότυπα, ιδίω στον τομέα των νέων τεχνολογιών και ε, συζητήσαμε και ότι πέραν των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να σημειωθεί πρόοδο πέρα από τις ε, κανονιστικές ρυθμιστικές αυτές συζητήσεις να σας πω ότι η Επίτροπος και ε, ο πρέσβης κατάφερε να κάνουν έναν απολογισμό για το που βρισκόμαστε. Κατέληξαν συζητήσεις μας αυτού του τρει τομεί που μόλι σα ανέφερα. Οι ρυθμιστικέ μα αρχέ πλέον βρίσκονται στη φάση του να προσδιορίσουν τι ακριβώ μπορεί να γίνει με ε, πλήρη σεβασμό των ε, εκάστοτε των αντίστοιχων ε, κανονιστικών πλαισίων των δύο πλευρών. Το δεύτερο θέμα αφορά την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Σε αυτό το θέμα είχαμε πολύ καλές συνομιλίες με τις ΙΠΑ για κάποια, θέματα, για το πώς μπορούν να ε, εφαρμοστούν οι κανόνες για τις επιδοτήσεις του ΠΟΕ, πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες ε, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις μεταφορές τεχνολογίας. Όπως ξέρετε, έχουμε υποβάλει μαζί με τις ΙΠΑ πρόταση στη Γενέβη για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια. Ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Δυστυχώ πρόοδο δεν μπορώ να σας πω ότι κάναμε. Το θέμα βρίσκεται στο αρμόδιο σώμα. Ε, συνεχίζονται οι συζητήσει και οι διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε υποβάλει την πρόταση και ελπίζουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε μια συμμετοχή των ΙΠΑ και σε αυτό το θέμα. Τέλος, είπατε κι εσείς το ζήτημα του, της έκθεσης της έρευνας 232 για τα οχήματα. Γνωρίζουμε ότι έγινε συζήτηση στο Λευκό Οίκο για αυτό το θέμα. Από αυτά που έχουμε καταλάβει δεν έχει οριστικοποιηθεί στάση από πλευράς ΙΠΑ για τον χρόνο ή τον, ε, το μέγεθος των ε, δασμών ε, σε σχέση με την έκθεση 232, όμως η Κομισιόν σε όλες τις επαφές ήταν ξεκάθαρη και με τον πρέσβη και με άλλους συνομιλητές μας ότι θα υπάρξει στεναρή απάντηση σε οποιαδήποτε έκθεση η οποία θα απειλήσει ή θα εφαρμόσει ποσοστώσεις ή δασμούς ε, σε εισαγωγές ευρωπαϊκών ε, αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Ε, ξέρετε ότι από τον Ιούλιο επεξεργαζόμαστε τον κατάλογο δασμών. Δημοσιεύουμε τα σχετικά στοιχεία μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο αλλά οποιαδήποτε κίνηση περιορισμού των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες δεν θα μείνει αναπάντητη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Με άλλα λόγια, θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση για ε, δασμούς όταν υπάρχει στον αέρα μια τέτοια έκθεση η οποία θέτει σε κίνδυνο τις ενωσιακές εξαγωγές και όλα αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν και από την ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει. Δεν υπάρχουν ε, άλλα, άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Αυτά που σας είπα δεν συζητούμε ούτε γεωργικούς δασμούς, ούτε σχετικές διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν κάποιοι, υπάρχει κάποια πρόοδος στα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΕ. Μπορώ να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες και πολύ ξεκάθαρη στάση από πλευρά μας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε διαπραγμάτευση υπό την απειλή διαφόρων εκθέσεων. Ιδίω όταν αυτό ε, ενδέχεται να επιφέρει και την επιβολή δασμών περίπτωση στην οποία, όπω ξεκαθαρίσαμε προ όλε τι πλευρέ, θα υπάρξει στεναρή απάντηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε. Τα επόμενα βήματα ε, σίγουρα θα περιλαμβάνουν κάποια πρόοδο και κάποια συνέχιση των συζητήσεων σε τεχνικό και ρυθμιστικό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και εκεί. Υπάρχει μια πιθανότητα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δύο πρώτων προέδρων στο περιθώριο του G20 που θα γίνει στο Buenos Aires και από την τεχνική πλευρά να σας πω ότι η Κομισιόν έχει ξεκινήσει την προετοιμασία δύο ε, ξεχωριστών ε, διαπραγματευτικών οδηγιών η μία για, τα βιομηχανικά, για τους βιομηχανικούς δασμούς αν τελικά ε, συμβεί κάτι τέτοιο και επιβληθούν τέτοια από τις ΗΠΑ και η άλλη οδηγία αφορά το ζήτημα της αξιολόγησης συμμόρφωσης, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που ρυθμιστικά μας έχει απασχολήσει και στο, ένα, είναι ένας τομέας στον οποίο χρειάζεται να συνεχιστούν οι διεθνείς συζητήσεις. Και σε αυτό το θέμα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε ε, οδηγίες διαπραγμάτευσης ε, σε εσά και στο Συμβούλιο. Σταματώ εδώ και βεβαίω, όπως είπα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες ερωτήσεις. Σχετικά με την εντολή. Το χρονοδιάγραμμα ποιο θα είναι. Θα συμμετάσχει το κοινοβούλιο μας στις συζητήσεις για την εντολή. Θα κάνω μια διάκριση ανάμεσα στην εντολή για την συμμόρφωση και το τεχνικό ζήτημα, γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δει η Επιτροπή όταν είναι έτοιμο το κείμενο τότε θα το υποβάλουμε στο Συμβούλιο. Και νομίζω ότι μπορεί να πάει αρκετά γρήγορα το θέμα λοιπόν το τεχνικό για την συμμόρφωση. Τώρα για το θέμα των δασμών, εκεί περιέχει και ένα πολιτικό στοιχείο. Οπότε οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολο να αρχίσουν χωρίς προηγουμένως να έχουμε ήδη κάποια άσκηση ώστε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Προς το παρόν δεν έχουμε καμιά αντίδραση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προς το παρόν μας λένε ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν μαζί μας εφόσον έχουν ε, τις 90 μέρες στο Κογκρέσο, οπότε θα φτάσουμε τον Μάρτιο. Και τότε θα μπορέσουμε δεχομένω να μιλήσουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε και να δούμε πού βρισκόμαστε ακριβώς. Και για να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχουμε καμία ιδέα και καμία πρόθεση να έχουμε ευρύτερες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Οι σκιώδη μας. Ο κύριος Ζαντό, Γιάννικ. Ευχαριστώ. Ιγνάσιο. Οι ευρωβουλευτές γενικά δεν είναι πονηροί και οι οικολόγοι είναι ακόμα λιγότερο από το μέσο όρο των ευρωβουλευτών. Και ειλικρινά μιλάω από μια στιγμή και μετά δεν καταλαβαίνω πια τίποτα στη διαδικασία που περιγράφεται. Ακούω μια λέξη που θέλετε να αποφύγετε να πείτε. Και αυτή είναι η εμπορική συμφωνία. Λέτε για τις βιομηχανικούς δασμούς. Διαπραγματευόμαστε για συμφωνίες συμμόρφωση και δεν ξέρω τι. Υπάρχει η Αμερικανική διαδικασία στο Κογκρέσο και φτάνουμε στα μέσα Ιανουαρίου. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα κατά πόσο θα διαπραγματευτούμε μία εμπορική συμφωνία. Ναι ή όχι. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, και πάλι σας είπα, έτσι δεν καταλαβαίνω και πολλά, είναι ότι αν διαπραγματευόμαστε για βιομηχανικούς δασμούς, πρόκειται για εμπορική συμφωνία. Κατάλαβα ότι δεν είναι συνολική συμφωνία, αλλά είναι μια διατλαντική εμπορική συμφωνία περιορισμένη στα βιομηχανικά ζητήματα συμμόρφωσης ίσως. Θα δούμε τι θα διαπραγματευτούμε και τι θα βγει από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αν είναι έτσι, ωραία, συμφωνούμε. Θα ζητήσετε εντολή, το είπατε, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα κάνει τη δικιά του τη δουλειά γνωμοδότησης, φαντάζομαι, για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά επί του παρόντος έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δεν είναι διαπραγμάτευση. Έγιναν δηλώσεις, τα πάμε, έγιναν δηλώσεις από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Καταλαβαίνω, jet lag και τα λοιπά. Το είπε όμως ότι εμείς θα προσφέρουμε περισσότερη σόγια τροποποιημένη, ε, περισσότερο αέριο σχιστόλιθου, τι γίνεται. Απαντάει έτσι σε, μια... σε κάτι που ζητούν οι Αμερικανοί ή ήταν το jet lag. Δεν ξέρω να μου το πείτε. Αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι πρόκειται για εμπορική συμφωνία που διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπραγματεύσεων και συζήτησης της εντολής για μια διατλαντική εμπορική συμφωνία. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ιγνάσιο, για την ενημέρωση. Γιατί χθες είχαμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συντονιστών ε, με την Επιτροπή για το θέμα αυτό, με την ίδια την Επίτροπο κιόλας. Και Γιάννικ είπε δεν είναι εμπορικέ διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας. Μιλάμε μόνο για τελωνιακούς δασμούς και μερικά βιομηχανικά προϊόντα με τη ΣΥΠΑ και μερικές ρυθμιστικές ε, σκοπιές που μόλις μας εξηγήθηκαν. Η ερώτησή μου προς τον Ιγνάθιο είναι η εξή. Αν είναι μόνο κάποια ρυθμιστικά αυτά που μας απασχολούν και μιλήσατε για τα φαρμακευτικά και τις ιατρικές συσκευέ. Ε, οι ρυθμιστικές ε, πτυχές της ΕΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι οι προδιαγραφές παρασκευής παραγωγής είναι διαφορετικές. Άρα γιατί μιλάμε. Άρα τελικά συζητάμε και πάλι για ρυθμιστικές πτυχές. Τι σημαίνει όλο αυτό. Η επόμενη ερώτηση είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το 232 και τα σχετικά προβλήματα. Εδώ μιλάμε για στοιχειωτικά ζητήματα, ζητήματα πολιτικής προστασίας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται και με την ε, ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Ποια είναι η θέση σας. Υπάρχει αβεβαιότητα για τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Πρόκειται να ληφθούν μέτρα προληπτικά από την αμερικανική πλευρά για να, πλευρά για να αποφύγουμε την ε, ανάληψη αντιπίνων από τον ΠΟΕ, η Αν Μαρή Μινέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω ερωτήσεις. Είμαι περίεργη. Η συνεργασία κρατιέται εκτός διαδικασίας υπάρχει, χρειάζεται μάλλον εντολή για τη συνεργασία, για την παράγραφο αυτή για τη συνεργασία. Ο κύριος Ντάρτμουθ, ευχαριστώ για τις διαπραγματεύσεις της εμπορικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα Είχαμε πριν λίγα χρόνια τέτοιες διαπραγματεύσει και είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και την Ολομέλεια. Θυμάμαι και όλε τι αντιδράσει τη τόσο γλαφριές και ζωηρέ του Πρόεδρου Σούλτ όταν ήταν ακόμα πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι είναι συναρπαστικό ότι υπάρχουν ε, διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΠΑ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικά επί εμπορίου το θέμα. Ε, μιλάμε για πολλού τομεί, αλλά όχι για το εμπόριο. Και Ξέρω κάποιον που επί 8 χρόνια ζούσε και εργαζόταν στη ΣΥΠΑ, ε, σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα, και γνώρισε πολλά για την Αμερικανική πολιτική και έλεγε ότι παραδοσιακά οι, παραδοσιακοί δημοκράτες ήταν το κόμμα του προστατευτισμού και οι ρεπουμπλικανοί ήταν ε, αυτοί του ελεύθερου εμπορίου. Με τον τωρινό πρόεδρο, οι ρεπουμπλικανοί έχουν γίνει το κόμμα του προστατευτισμού. Και δεν θα αναφέρω καν και το όνομά του, διότι φαίνεται ότι θα χάσουμε λίγο τον μπούσουλα και δεν θα σκεφτόμαστε πια το εμπόριο. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει ε, με το ελεύθερο εμπόριο και ο κυβερνήτης του Χάιο είναι ο ε, αυτός πρωτοστατεί στον προστατευτισμό τη ε, ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης. Το θέμα είναι να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικέ εμπορικές δραματεύσεις είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουμε θέματα όπω τα γεωργικά και τόσα άλλα. Εκτός λοιπόν αν γνωρίζετε κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε, θα ήθελα να μας πείτε. Ε, και αυτή είναι η ερώτησή μου. Οι εμπορικέ αυτέ διαπραγματεύσει είναι εμπορικέ ή όχι. Απλώ καθέστε και συζητάτε για κάποιου ε, αδιάφορου τομεί εμπορίου. Εγκνάσιο και εγώ από την πλευρά μου. Οι δασμοί για τα εμπορικά αγαθά χωρίς τα αυτοκίνητα δεν μας ε, βοηθά χωρίς συγκεκριμένους αριθμούς. Ποιος όγκος συναλλαγών καλύπτεται από αυτά τα προϊόντα και ποιες ε, τελωνιακές γραμμές. 7%, 15%, 80% γιατί μιλάμε. Και αυτά θα γίνονταν αποδεκτά από τον ΠΟΕ Και επίσης δεν μου αρέσει καθόλου ο αποκλεισμό των αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια μόνιμη απειλή. Θα υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθούν δασμοί για τα αυτοκίνητα. Βάσει της νομοθεσίας 232 που μας έχει μείνει από τον ψυχροπόλεμο από το 1962 Είναι μια απειλή διαρκείας αυτή. Είναι σοφό να έχουμε συμφωνία που να δέχεται αυτή την ε, διαρκή απειλή. Ναι. une petite question supplémentaire. Μια μικρή ερωτησούλα, εξτρά. Ε, Ιγνάσιο, αναφέρατε τις προθεσμίες 90 ε, ημέρες, μέσα Ιανουαρίου και το καθεξής. Ε, από αυτά που καταλαβαίνω από την Αμερικανική διαδικασία, η κυβέρνηση θα πρέπει να δημοσιοποιήσει 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ε, των μέσων Ιανουαρίου την ε, διαπραγματευτική της πρόθεση. Δηλαδή, όλοι θα γνωρίζουμε τι θα θέλουν οι Αμερικανοί περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η προθεσμία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω στην επίσημη και τυπική της συνεννόηση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Ιγνάθιο, για όλες αυτές τις επεξηγήσεις. Έχω την εξή ερώτηση. Είτε ονομάζεται εμπορική συμφωνία, είτε όχι. Διαπραγματευόμαστε όμως για κάτι που έχει να κάνει με το εμπόριο, οπότε συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο εδώ Ζαντό. Όπως και να το ονομάζουμε όμως. Ετοιμάζουμε ένα πλαίσιο σχέσεων που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όμως ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε υποχώρησαν από τη Συμφωνία των Παρισίων και ακριβώς η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με τα βιομηχανικά αγαθά. Έπειτα, το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξης. γιατί δεν είναι σημαντικό όταν πρόκειται για ανταλλαγή βιομηχανικών προϊόντων όταν πρόκειται για τη γεωργία και τις υπηρεσίες είναι και εδώ δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μία συμφωνία καθαρά για βιομηχανικά προϊόντα θέτει σε κίνδυνο όλη την πρόοδο που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα όσον αφορά τις αρχές μας που πρέπει ακριβώς να συνάδει με οποιαδήποτε νέα εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με το ερώτημα του κύριου Ζαντό. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν αποσκοπούμε στο να διαπραγματευτούμε για πολλούς λόγους μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μπορώ να σας δώσω τους λόγους, είναι πολλοί. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανταποκριθούν σε πολλές από τις προτεραιότητες που θα θέσουμε εμείς και σε περίπτωση ε, εμπορικής σύγκρουσης λόγω αυτής της πιθανότητας λοιπόν αποφασίσαμε και οι δύο πλευρές, οι δύο πλευρές να περιορίσουμε τη συζήτηση στο ζήτημα των βιομηχανικών δασμών. Βεβαίως η συζήτηση αυτή αφορά το εμπόριο, αλλά δεν είναι μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία, μια ολοκληρωμένη εμπορική διαπραγμάτευση. Επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα των βιομηχανικών δασμών. Για το ε, LNG και τη σόγια, τα δύο θέματα που αναφέρατε. Ξέρετε ότι στη σόγια ε, δεν υπάρχει δέσμευση να αλλάξουμε την πολιτική που ακολουθούμε, απλά επαληθεύσαμε ότι για μια σειρά λόγους υπάρχουν αυξημένες εισαγωγές σόγιας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ζήτημα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι υπάρχει ε, συμφέρον και επιθυμία να ε, συνεχιστούν οι συζητήσεις για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και αν ληφθεί κάποια δράση αυτή θα πρέπει να προέλθει από τις ΙΠΑ, διότι οι ΙΠΑ είναι εκείνες που αυτή τη στιγμή ε, εφαρμόζουν περιορισμούς όσον αφορά τις εξαγωγές LNG. Να απαντήσω και για το ζήτημα των 30 ημερών. Η αρχή πρόθεση του εμπορίου δεν λέει ότι η κυβέρνηση αυτή ε, πρέπει ε, μετά τις 90 μέρες εντός 30 ημερών να ζητήσει εντολή διαπραγμάτευσης. Λέει ότι 30 μέρες πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης θα πρέπει αυτή η κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοποίηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή αφότου ε, παρέλθουν αυτές οι 90 ε, ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ΙΠΑ δεν είναι καθόλου υποχρεωμένε να έρθουν σε επαφέ μαζί μα για να δούμε ποια θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση. Εμεί ελπίζουμε ότι θα το κάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαβούλευση των 90 ημερών στο Κογκρέσο και αφού αυτέ εκπνεύσουν θα έρθουν, ελπίζουμε, οι ΙΠΑ σε εμά και να μας πούν ότι θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις μαζί σας για, ε, με απότερο σκοπό την κατάργηση των ε, βιομηχανικών δασμών. Αυτό και μόνο αυτό. Για τα ε, ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Σόλτς. Γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι προτού περάσουμε σε πιο λεπτομερείς συζητήσεις με, τους, με τις ρυθμιστικές αρχές στην Ουάσινγκτον... Ε, δημοσιεύσαμε και κοινοποιήσαμε σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποια, ε, ποια θέματα θεωρούμε ότι ενδείκνυνται ε, για εμβάθυνση και της συνεργασίας και προόδο σε ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου. Ξέρετε ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις καλές πρακτικές μεταποίησης, αλλά τη συμφωνία αφορά αυτή τη στιγμή μόνο τα φαρμακευτικά προϊόντα. Βεβαίω, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και τη δυνατότητα να διευρυνθεί ε, στα εμβόλια και τα κτηνιατρικά φάρμακα και αυτά είναι τα θέματα που συζητούν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εδώ υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα από τα θέματα είναι πώς θα είναι συμβατά τα συστήματα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, πώς θα ταιριάζουν, πώς θα είναι διαλειτουργικά και αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε καταλήξει με τη ρυθμιστική αρχή τον είπα ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις, ότι μπορούν να γίνουν συζητήσεις Ξαναλέω, μιλώ για την ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και το άλλο ζήτημα που έχουμε συζητήσει είναι τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει βήματα προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει σε μια πολυμερή συμφωνία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δηλαδή, να κάνουμε τα ίδια που έχουν ήδη γίνει στον τομέα των φαρμάκων, προκειμένου να αποφεύγονται ε, η διπλή έλεγχη, αν θέλετε. Αυτά είναι τα θέματα που έχουμε συζητήσει σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών και στα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σημειωθεί προόδος βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Θα επανέλθω και στο ζήτημα του 232, αλλά θέλω πρώτα να συνεχίσω λίγο με τα ρυθμιστικά ζητήματα. Εξετάζοντας τα ζητήματα που έχουμε ε, συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει μόνο ένα θέμα στο οποίο έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο και να ζητήσουμε ε, κατευθύνει γραμμέ διαπραγμάτευση. Και αυτό αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωση. Και ο λόγο είναι ότι αυτά που έχουν συζητηθεί θα απαιτήσουν σύναψη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών μιας διεθνούς συμφωνίας και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει προηγηθεί πρώτα ε, εντολή διαπραγμάτευσης από το Συμβούλιο. Γι' αυτό και ε, εξετάζουμε τη μορφή που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εντολή διαπραγμάτευση. Βεβαίως το ότι είναι αναγκαία αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουμε κρυφά. Αντίθετα, η πρόθεσή μας είναι να είμαστε απόλυτα διαφανείς γύρω από τα ρυθμιστικά ζητήματα που συζητούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ξεκαθαρίζοντας πάντοτε ότι δεν πρόκειται να λάβουμε καμία δράση που θα επιφέρει αλλαγή του ρυθμιστικού μας πλαισίου. Απλώς διερευνούμε διάφορες δυνατότητες για την ενίσχυση της ε, συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών μας αρχών. Και ταυτόχρονα ξεκαθαρίζουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από ρυθμιστικά ζητήματα θα πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρη από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τους βιομηχανικούς δασμούς. Γιατί θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η συζήτηση γύρω από τα ρυθμιστικά ζητήματα δεν θα μπερδευτεί με ε, ζητήματα εμπορικά, βιομηχανικών δασμών κτλ. κτλ. Θεωρούμε ότι αυτά τα δύο θέματα πρέπει να εξεταστούν αυτόνομα. Για το άλλο ερώτημα, η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι ε, ε, θα επανέλθουμε σε μια διαδικασία ε, διαπραγμάτευση ολοκληρωμένη εμπορική ε, συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, ακριβώ γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητε ισορροπίε. Για τα ζητήματα που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από τη διαπραγμάτευση σχετικά με την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών. Η ΙΠΑ φαίνεται ότι έχουν άλλη άποψη και γι' αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν οπωσδήποτε προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Μια συμφωνία που θα καταργεί ε, του δασμού σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά όχι τα γεωργικά προϊόντα, κατά τη γνώμη μα είναι κάτι εφικτό από άποψη συμφόρφωση με το άρθρο 24 της ΓΚΑΤ ε, θα καλύπτει το εμπόριο κατά 95%, τις εμπορικές συναλλαγές δηλαδή κατά 95%, δεν τα θυμάμαι και ακριβώς απ' ε, έξω, αλλά πάντως πάνω από 90% των εμπορικών συναλλαγών θα καλύπτονται από μια τέτοια συμφωνία και από την σκοπιά του ΠΟΕ θεωρούμε ότι αυτό θα είναι μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως εφικτή σχετικά με την ε, συμμόρφωσή της με το άρθρο 24. Φυσικά ε, μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα επιβατικά οχήματα είναι μια λίγο διαφορετική υπόθεση γιατί υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ σε κάθε περίπτωση ε, θα συζητηθούν ξεκάθαρα όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά και υπό το πρίσμα της ε, συμβατότητας με τους κανόνες του ΠΟΕ ώστε να μην καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι ε, παράτυπο. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες στην αυτοκινημιομηχανία. Μπορούμε να συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα ε, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλα αυτά είναι ανοιχτά προς συζήτηση. Νομίζω ότι έχω ξεκαθαρίσει ότι αν δεχθούμε απειλή όσον αφορά την επιβολή ποσοστώσεων ή δασμών στα αυτοκίνητα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε καν την διαπραγμάτευση. Τι θα γίνει αν έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, βεβαίω και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη εξέλιξή τη θα επιβληθούν τέτοιοι δασμοί. Μα είναι σαφέ, θα ανασταλούν διαπραγματεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε σε συμφωνία για του δασμού με τη ΣΥΠΑ υπό την απειλή επιβολή δασμολογικών μέτρων. Και έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, δεν ε, είμαστε πρόθυμοι να συμφωνήσουμε σε ποσοστώσεις για ε, τα αυτοκίνητα. Και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων μας υπό τον ΠΟΕ. Για τον χάλιβα και το αλουμίνιο η Επίτροπος Μάλστρομ το έχει θέσει σε όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που είχε και με τον πρέσβη, τον ομόλογό της. Έχουν γίνει προσπάθειες να εξευρεθεί λύση και για το ζήτημα των, της επιβολής δασμών και των αντίμετρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει κάποια προσφορά από τις ΗΠΑ που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Μας έχουν πει ότι ίσως οι ΗΠΑ μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ποσοστό σε αντίδασμών. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όπως λέει και ο ΠΟΕ οι ποσοστώσει είναι παράνομες και από πολλέ απόψεις είναι και χειρότερες από τους δασμούς, γι' αυτό και δεν αποτελούν επιλογή για εμάς. Γενικά ε, δεν φαίνεται να υπάρχουν καλές δυνατότητες επίλυσης αυτή τη στιγμή του ζητήματος. Φυσικά η Μακουλάδα έκανε τη μάλλον πιο δύσκολη ερώτηση προς το τέλος πρέπει να καταλάβουμε το ειδικό περιβάλλον στο οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται σε ένα πλαίσιο όπου προσπαθούμε να αποφύγουμε μεγάλη κλίμακα εμπορική σύγκρουση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα δείτε υπό το πρίσμα του τι, να, τι μπορεί να γίνει για να αποφευθεί μια τέτοια εμπορική σύγκρουση. Μία από τι απαντήσει που δίνουμε είναι ότι μιλάμε για μια διαπραγμάτευση πολύ περιορισμένη που θα αφορά μόνο τους βιομηχανικού δεσμού, για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και δεν πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν κατάλληλο ε, ή σωστό να πω ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη ή το άρθρο 23. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση όπως έχω πει ήδη πολλές φορές είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αν θέλετε το περιβάλλον στο οποίο ε, λαμβάνουν χώρα αυτές οι συζητήσεις και όλα αυτά συνεκτιμώνται δεόντως από εμάς. Καλώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ευχόμαστε καλή, ευχόμαστε καλή τύχη. Το τελευταίο θα πρέπει να είναι η ανταλλαγή απόψεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και ιδίω ε, για τη μελλοντική εμπορική και οικονομική εταιρική σχέση. Όμως, όμως, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι ο χρόνος που έχει περάσει και μας μένουν μόνο 10 λεπτά. Δεύτερον, ο εισηγητής μας δεν είναι διαθέσιμος. Και τρίτο, αυτό βέβαια είναι δικό μου, θα θέλαμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως είπαν ότι δεν μπορούν να έρθουν. Το έβαλα στην ημερήσια διάταξη γιατί σεβόμενος βέβαια πάντα τις αρμοδιότητες της κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, είναι η ΑΦΚΟ και άλλες επιτροπές υπεύθυνε για την συμφωνία και την αποχώρηση. Τώρα όμως πρόκειται για την δήλωση όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου που έρχεται τα γενεθλιά μου. Επί τη ευκαιρία, λέει ο Πρόεδρος. Θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει βάση για συζήτηση όσον αφορά το εμπορικό σκέλος τη συμφωνίας και των μελλοντικών σχέσεων. Όπως όμως σας είπα και νωρίτερα, η ομολογή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διαπραγματευτική ομάδα, δεν είναι εδώ. Και επειδή δεν έχουμε και αρκετό χρόνο, θα πρότεινα να αναβληθεί η συζήτηση για αυτό το θέμα. Βέβαια, αν έχετε σχόλια, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Συμφωνώ με την αναβολή βεβαίω. Αλλά θέσατε και τη μία και μόνη ερώτηση που θέλω να θέσω και εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν είχε έρθει. Το τμήμα των πολιτικών δηλώσεων και βάσει και τη δική σα επιχειρηματολογία δεν είναι το τμήμα που αφορά και το εμπόριο και θα έπρεπε να μα απασχολήσει ω διαπραγματευτική εντολή. Πού είναι αυτή η διαπραγματευτική εντολή και τι καθεστώ θα έχει. Διότι αν είναι μια γενική δήλωση, ε, ποιο είναι το νόημα. Αλλιώ πώ θα υπάρξει αρχή των διαπραγματεύσεων. Πράγματι. εξ όσων γνωρίζω δεν είναι νομικό δεσμευτικό κείμενο. Θα καλύπτει και άλλες πτυχές από τις εμπορικές, όπως φαντάστηκα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει εντολή για πραγματικές διαπραγματεύσει. Χέλμουτ. Ευχαριστώ να τα αναβάλουμε. Αλλά ως προς το πρόγραμμα να προετοιμαστούμε διότι το αργότερο μετά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, εάν δεν γίνει έκτακτο το επόμενο Σαββατοκυριακό, για να καταλήξουμε σε μια θέση εμείς ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είμαστε υπεύθυνοι να σκεφτούμε τις μελλοντικές μας σχέσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε κατά λεπτό τι προκλήσει και τι θέλουμε στο μέλλον. Οικονομικό, εμπορικό κτλ. Τη συνεργασία μα. Μήπω πρέπει να συζητήσουμε έτσι κι αλλιώ για να επηρεάσουμε την εντολή που μπορεί να δοθεί για τι διαπραγματεύσει find Μη βρεθούμε στριμωγμένοι να έχουμε σκεφτεί με υπεύθυνο τρόπο ούτω ή άλλω την μελλοντική πορεία. Κύριο Συμφωνώ με την αναβολή. Έχω κάτι διαδικαστικό να ρωτήσω. Υπάρχει πιθανότητα η Επιτροπή μας να απαιτήσει από την Επιτροπή να στείλει εκπρόσωπο. Μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε πράσινο φως για, για να το... Δεν έχουμε δικαίωμα να τους υποχρεώσουμε. Λοιπόν, πάμε στο 29, διάφορα, το αγαπημένο μου, κανένα. Επόμενη συνεδρία 3 Δεκεμβρίου. Τέλος.